Colleagues, good afternoon. Καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Ξεκινάει η συνεδρίασή μας. Έχετε την ημέρη σε διάταξη ενώπιόν σας. Ε, την δέχεστε, έχετε κάποια παρατήρηση. Ωραία. Πάμε στο θέμα CARS 2020, εξέταση των τροπολογιών. Ο κύριος Βλάσεκ ζητά συγγνώμη, αλλά Ο κύριος Μπραντμπορη. Ναι, μου έχει δώσει μία δήλωση την οποία θα ήθελε να σας παρουσιάσει. Ζητά συγγνώμη για το γεγονός ότι δεν μπόρεσε να είναι παρόν στις Βρυξέλλες σήμερα. Για τη γνωμοδότηση, ο κύριος Βλάσεκ χαιρετίζει το θετικό έργο των σχεδόν εισηγητών και των άλλων συναδέλφων που έχει συμβάλει ιδιαίτερα στη συζήτηση και εν γέννη οι τροπολογίες οι οποίες έχουν κατατεθεί δείχνουν κάθε θέληση να ενισχυθεί η αντιαγωνιστικότητα και η απόδοση τη ευρωπαϊκής Αυτοκινητοβιομηχανία και επίσης να εξασφαλίσουν τις θέσεις απασχόλησης οι οποίες κινδυνεύουν από τη μείωση του όγκου πωλήσεων αυτοκινήτων. Επίσης, χαιρετίζει τι τροπολογίες που ζητούν μια πιο συνεκτική προσέγγιση της Κομισιόν για την αυτοκινητοβιομηχανία που βασίζονται σε λεπτομερή αξιολόγηση των νομοθετικών προτάσεων, όπως παραδείγματος χάρη αναφέρεται στις τροπολογίες 41-42. 42 Υπογραμμίζει την ανάγκη να υπάρχει τεχνολογικά ουδέτερη έρευνα και καινοτομία για την αυτοκινητοβιομηχανία με στόχο την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας και επίσης χαίρεται για αυτά τα οποία αναφέρονται σε σχέση με τη δημιουργία μιας εναλλακτική υποδομής και την εναρμόνιση των τεχνικών προτύπων που καλύπτεται από την τροπολογία 31. Η τροπολογία 7 αφορά τον όγκο πωλήσεων και τονίζει το γεγονός ότι αλλάζει η συμπεριφορά των καταναλωτών. Και τέλος, Υπάρχει μια σειρά τροπολογιών που σύμφωνα με τον εισηγητή απομακρύνονται πάρα πολύ από τον αρχικό στόχο της έκθεσης διατήρηση θέσεων απασχόλησης, δηλαδή και ανταγωνιστικότητα και κύριο Βλάσακ θέλει να τονίσει ιδιαίτερα την ανάγκη ότι δεν πρέπει να παρέμβουμε στον τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνουν τους στόχους διοξιδίου του άνθρακος η αυτοκινητοβιομηχανίας. Αν εφαρμόσουμε υποχρεωτικές κατευθύνσεις, παραγωγός χάρη, όρια σε ό,τι αφορά την έρευνα για την αεροδυναμική κτλ. Η κατασκευή κινητήρων, ελαστικών, εναλλακτικές τεχνολογίες, χρήση ε, καυσίμων κτλ. Όλα αυτά μπορούν να τροχοπεδίσουν τη διαδικασία μείωσης των εκπομπών διοξιδίου του άτομου. Αυτά είναι τα συμπεράσματα του κ. Βλάσακ. Ευχαριστώ. Που παρουσιάσετε την άποψη του κ. Βλάσακ. Ο Μάτιου για τον κύριο Φέρμπερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και ο κύριος Φέρμπερ δυστυχώς δεν μπορεί να είναι εδώ παρόν, είναι στο Μόναχο. Αλλά θεωρεί ότι εν γέννη η έκθεση του εισηγητή είναι ιδιαίτερα θετική Έχει καταθέσει μονάχα τέσσερις τροπολογίες ο κύριος Φέρμπερ, όπου φυσικά θέλει και αυτός να υπογραμμίσει την πρόταση αυτή ότι μέσα από την έρευνα και την καινοτομία στον τομέα αυτό θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη υποστήριξη, ότι θα πρέπει να εντοπίσουμε εκεί που υπάρχουν προβλήματα και ασφάλματα, το γεγονός ότι υπάρχει μια υποδομή η οποία δεν έχει συμπληρωθεί πλήρως και αυτό αφορά κυρίως τις εναλλακτικέ μορφές προώθησης των οχημάτων, αλλά σημαίνει επίσης ότι και σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να υπάρξει μια μεγαλύτερη εναρμόνιση και τυποποίηση για όλα τα πρότυπα, γιατί αλλιώς ελοχεύει ο κίνδυνος ότι δεν θα μπορέσει να υπάρξει μια αρμονική εξέλιξη στον χώρο της αγοράς, επειδή θα υπάρχει απαραίτητη διαλειτουργικότητα μεταξύ των οχημάτων και της υποδομές. Είναι ένα πρόβλημα που γνωρίζουμε και από άλλους τρόπους μεταφοράς. Τονίζει επίσης ότι δεν πρέπει να είμαστε περιοριστικοί, αλλά θα πρέπει να προσπαθήσουμε να είμαστε προορατικοί και να υποστηρίζουμε. Αλλά φυσικά δεν μπορούμε να απογυμνώσουμε τις επιχειρήσεις από τη δική τους ευθύνη που είναι να επιτύχουν τους στόχους αυτούς όπως έχει τονιστεί ιδιαίτερα από την ομάδα υψηλού επίπεδου σε διάφορες ε, ευκαιρίες. Θα πρέπει όλοι αυτοί οι οποίοι εμπλέκονται να αναλάβουν την ευθύνη να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι και όχι μονάχα ο τελικός κατασκευαστής. Ελπίζουμε επίσης ότι στο μέλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορέσει να έχει ένα εμπορικό και κατασκευαστικό μέλλον για την αυτοκίνητο βιομηχανία Πρέπει όμως να βελτιωθεί η ανταγωνιστική θέση της Ευρώπης για τα θέματα αυτά με μέτρα τα οποία δεν θα έχουν περιοριστικό χαρακτήρα. Πιστεύουμε ότι είναι η σωστή κατεύθυνση, είναι η σωστή οι στόχοι οι οποίοι έχουν τεθεί και τονίζει ιδιαίτερα ότι θα πρέπει να εντοπίσουμε ιδιαίτερα τα προβλήματα και να τα αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε η κυρία Λζαμπάλα έρχεται στο Κοινοβούλιο και μου ζήτησε να την αντικαταστήσω. Θα είμαι σύντομος, διότι λυπούμεθα ιδιαίτερα που θα, ε, που θα πρέπει να ομολογήσουμε ότι ο εισηγητής δεν δέχτηκε τις τροπολογίες μας, τις περισσότερες τουλάχιστον, και δεν έχουμε την δυνατότητα, δεν είχαμε τη δυνατότητα να το συζητήσουμε με τον εισηγητή. Δεν υπήρχε καμία οργάνωση ε, συνάντησης ε, μεταξύ των σκιωδών εισηγητών, επομένως δεν προτάθηκε καμία συμβαστική πρόταση. Ε, δεν είναι ο σωστός τρόπος δουλειάς, πιστεύουμε, και θα δούμε πώς θα τελειώσουν στην ψηφοφορία τα πράγματα. Τέλος πάντων, εμείς θέλαμε να υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα στους πυλώνες του προγράμματος δράσης, στηριζόμενη σε ε, μια βιώσιμη δράση και στις δυνατότητες ανάπτυξης και όσον αφορά τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, θέλουμε να είμαστε συνεπείς με την θέση που θέτει στο Κοινοβούλιο για τα αυτοκίνητα και για την οδηγία, ε, τον κανονισμό, συγγνώμη, για το για τις εκπομπές ε, διοξιδίου του άνθρακα που βάζει σαν ε, στόχο το 2017 όσον αφορά τις εκπομπές ε, διοξιδίου του άνθρακα των αυτοκινήτων. Αυτά είναι τα επιχειρήματά μας. Αυτά δεν δυστυχώς λήφθησαν υπόψη. Λυπούμεθα γι' αυτό. Σας ευχαριστούμε πάντως και ελπίζουμε ότι θα προσαρμοστεί και, η, και ο κατάλογος των ψηφοφοριών ανάλογα. Η κυρία Μάισερ.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 <laughs> Ε, Α, 2017. Λοιπόν, εκεί έχει τεθεί ε, σαν όριο ε, για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα 68 έως 78 γραμμάρια ένα χιλιόμετρο. Αυτή είναι η τροπολογία 23 του κύριου Τέλερ και 27 του εισηγητή από την ομάδα των σοσιαλιστών. Επίσης, ε, μέσα στα πλαίσια της καταπολέμησης ε, των κλιματολογικών αλλαγών, υπενθυμίζει ότι η βιομηχανία μας ε, περνάει μια κρίση και επομένως δεν θα πρέπει να υποβληθεί σε περαιτέρω κυρώσεις. Επίσης, ζητάει ξεχωριστή ψηφοφορία για την ε, τροπολογία 14 της ε, έκθεσης του κ. Βλάζακα. Ε, επιβεβαιώνεται επομένως εδώ η θέση της όσον αφορά την οδική ασφάλεια. Όμως δεν υποστηρίζει, υποστηρίζει το πρώτο κομμάτι της τροπολογίας αυτής, αλλά όχι το δεύτερο, που όσον αφορά τα όρια ταχύτητας. Ευχαριστώ κύριε Μάισνερ. Τόσο καλά περί... σχεδόν σαν τα δικά μου. Κύριε... Κράμερ, θέλετε να πείτε κάτι κι εσείς. Ε, ευχαριστώ, Μάικλ. Η Κομισιό. Η κυρία Κοξόβα. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις τροπολογίες και για τη δουλειά που έχει γίνει. Δεν Έχουμε συγκεκριμένη παρατήρηση ή σχόλιο μέχρι στιγμής. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας αυτό για την οικονομική, την οικονομική κατάσταση, την οικονομική κρίση και να προσαρμοστεί η έκθεση. Η, η κατάσταση της αυτοκινητοβιομηχανίας εξελίσσεται καθημερινά και οι πρόσφατες εξελίξεις είναι λίγο πιο αισιόδοξε. Δηλαδή υπάρχει μια κάποια ελπίδα και δεν χρειάζεται να είμαστε τόσο σκληροί. Θέλεις να πεις τίποτα Φίλιππ. Μήπως θα μπορούσε να περάσεις ε, το μήνυμα στον εισηγητή, γιατί με ανησυχεί το γεγονός ότι δεν υπήρξε συνάντηση με τους κοιόδης. Πες του το, γιατί δεν είναι ο κατάλληλος τρόπος για να δουλέψουμε, αλλά τέλος πάντων αυτή είναι η κατάσταση τώρα. Αύριο ψηφίζουμε. Πάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Ευχαριστώ πάρα πολύ φίλοι που ε, κάλυψε το κενό. Επόμενο σημείο, επιτήρηση εξωτερικών θαλασσίων συνόρων. Η έκθεση της κυρίας Γκρίσμπεκ. Α, μόλις έφτασε... Έφτασε από τη Γαλλία ή εσύ πάλι είσαι. Πάλι εγώ στα γαλλικά. Πάρα πολύ ωραία. Δεύτερο μάθημα. Η κυρία Μάισνερ για να αντικαταστήσει την κυρία Γκρίσμπεκ για τα εξωτερικά θαλάσσια σύνορα. Πρόκειται για ένα κείμενο το οποίο αφορά τα εξωτερικά θαλάσσια σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το οποίο αφορά την... και ανήκει πάνω στη διακαιδοσία της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Με δυσκολία όσο και να το, να το, να το ε, ε, δούμε το θέμα από, την, από άλλη γωνιά, τέλος πάντων πρέπει να πούμε ότι ε, δεν αντιμετωπίζεται σωστά η κατάσταση. Εδώ θα πρέπει να δούμε δύο πτυχές ε, με τις οποίες εστίασε την ε, εργασία της ε, η κυρία Γκρίσμπεκ. Το ένα είναι η εκπαίδευση των ε, υπευθύνων για την, για την διάσωση των ανθρώπων που κινδυνεύουν. Και δεύτερον είναι η θαλάσσια επίβλεψη τέλο πάντων. 17 τροπολογίες υποβλήθηκαν, η κυρία Γκρίσμπεκ υποστηρίζει όλες εκτός από 6. του κυρίου Ντανιέλη, στις 19 και 20 του κυρία Τέιλορ και την τροπολογία 14 Φιντάνσα των Πρασίνων. Χωρίς να μπούμε σε λεπτομέρειες, δεν υποστηρίζει η κυρία Γκρίσμπεκ τις τροπολογίες αυτές, γιατί δεν αφορούν ε, κάποια σημεία ε, που την ενδιαφέρουν άμεσα ή δεν υπάρχουν κάποιες, δεν καλύπτονται κάποιες πτυχές όσον αφορά την επιθεώρηση των πλοίων. Αυτά για τις ε, τροπολογίες 17-18-19 και η 10 που καταργείται μια, ε, ένας ορισμός. Αυτά. Okay. I take it, Mr. Grosch, again. Ο κύριος Γκρόσο για τους ΕΛΚΑ. Και... Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο κύριος Φιντάντσα δεν μπορούσε να είναι εδώ παρόν. Αλλά εν γέννη χαιρετίζει την έκθεση του εισηγητή μας, τονίζει ότι τα κυριότερα σημεία, ιδίως στο θέμα της εκπαίδευσης, αναλύονται σωστά, ώστε να υπάρχει σωστή δυνατότητα εξοπλισμού και όλα αυτά τα θέματα θα πρέπει να λυθούν υπόψη μέσα στα προλέσια της έρευνας και της ανάπτυξης, όπως είναι παραγωγός το πρόγραμμα Horizon 2020. Και είναι σημαντικό επίσης να υπάρξει μια ανταλλαγή πληροφοριών με καλύτερο τρόπο και επίσης έχει καταθέσει μια τροπολογία με στόχο όχι να περιορίσει τις απόψεις της Επιτροπής Μεταφορών, αλλά να μπορέσει να βελτιώσει την προσθέμενη αξία που μπορεί να προέλθει από την ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων, όπως ε, ανέφερε και η Γκεζίνε. Ο στόχος λοιπόν είναι τα θέματα αυτά να ολοκληρωθούν εδώ και όχι να παραπενθούν σε άλλες επιτροπές όπως είναι η ΛΥΜΠΑ. Ευχαριστώ. Κύριε Αλκαντράου, για τον κύριο Δανέλη. Στα ελληνικά φαντάζομαι. Όχι, όχι στα ελληνικά λέει ο κύριος Αλκαντράου. Θα είστε ευγνώμων ίσως γι' αυτό η ομάδα μας και ο σκιώδης εισηγητής μας θέλουν να ευχαριστήσουμε τον εισηγητή για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε. Ο κύριος στόχος της απόφασης του Συμβουλίου του 2010 και του προτινόμενου κανονισμού που έχουμε τώρα ενώπιόν μας ήταν να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες οι οποίες υπήρχαν για τις θαλάσσιες ενέργειες της Frontex. Τα κράτη-μέλη και η ΜΚΟ είχαν εκφράσει ανησυχία σε ό,τι αφορά τα θέματα προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια αυτών των επιχειρήσεων στην ε, στα διεθνή ύδατα. Η πρόταση αυτή, ιδίω με το άρθρο 4 για τα θεμελιώδη δικαιώματα, αντιμετωπίζει κάποιε από αυτέ τι ανησυχίε και το κείμενο του εισηγητή και οι τροπολογίε που κατετέθηκαν βελτιώνουν το κείμενο αυτό, δίνουν περαιτέρω ρήτρε για ιατρική βοήθεια και υποχρεώσει για ασφάλεια κατά τη διάρκεια αυτών των ναυτικών επιχειρήσεων. Χρειάζεται όμω περισσότερη προσοχή σε ό,τι αφορά τι επιχειρησιακέ πλευρέ τη θαλάσσια εποπτεία. Το σημαντικό είναι να μπορέσουν να εφαρμόζονται σωστέ αρχέ αλλά τελικά η αρχή για το πώς θα πρέπει να λαμβάνεται να γίνονται αυτά στην πράξη θα πρέπει να παραμένει στην κρίση του πληρώματος του σκάφους. Αυτό το οποίο χρειάζεται ένα κοινό πλαίσιο το οποίο προστατεύει τα θεμελιώδη δικαιώματα και εξασφαλίζει ότι υπάρχει πλήρη συμμετοχή των κρατών μελών και οδηγεί σε μια ενιαία ερμηνεία του διεθνούς δικαίου. Αυτά λοιπόν και μπορούμε να συμφωνήσουμε με τη γραμμή του εισηγητή και ευχαριστούμε πολύ τον εισηγητή για τη συνεργασία του. Ευχαριστώ πολύ, λέει και ο πρόεδρος. Μάικλ, θα λάβει τον λόγο για τα θέματα αυτά. Κράμερ. Και για το δικό μα συζητή, ο οποίος δεν είναι παρό, είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία για τα θέματα της έκθεσης Γκρίσπαχ. Κάναμε μια τροπολογία σε ό,τι αφορά τους πρόσφυγες. Θεωρώ ότι δεν είναι δυνατό ένας ε, πρόσφυγας να μην αντιμετωπίζεται και να μην ασχολούνται τα πλοία με αυτόν. Θα πρέπει τουλάχιστον να συλλέγεται και να του δίδονται τρόφιμα και κουβέρτες. Το αν είναι νόμιμο ή όχι, αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί όταν αποβιβαστεί στην ξηρά. Δεν θα πρέπει λοιπόν να αγνοούνται οι πρόσφυγε στη θάλασσα, κάτι το οποίο έχει γίνει πολλέ φορέ. Θα πρέπει να υπάρχει μια πιο προσεκτική αντιμετώπιση από ό,τι μέχρι στιγμή έχει γίνει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Από την Κομισιόν η κυρία Χίλη. Thank you and good to... Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα σε όλους. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις προτινόμενες τροπολογίες. Έχουμε δύο γενικά σχόλια, αν μου επιτρέπετε. Ένα πρώτο σχόλιο το οποίο ήδη είχα εκφράσει παλιότερα όταν ε, παρουσίασε το σχέδιο γνωμοδότησης η και όσον αφορά τις τροπολογίες για τους εξοπλισμούς και τις προμήθειες πίτων σκαφών είναι μια τροπολογία σημαντική για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας και για την ασφάλεια των ανθρώπων που διασώζονται βεβαίως αλλά Πιστεύουμε επίσης ότι θα πρέπει να θεωρηθεί ως ένας κανονισμός πλαίσιο, για ένα κοινό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις στη θάλασσα και ότι λεπτομέρειες των διατάξεων όσον αφορά κουβέρτες, τρόφιμα κτλ. θα πρέπει να φεθούν στην κρίση των ομάδων που συμμετέχουν στην επιχείρηση. Θα ήθελα να τονίσω μια αναφορά που γίνεται στην τροπολογία 14 σε διμερείς συμφωνίες. Αυτό, αυτή αφορά τις, ε, τα θεμελιώδη δικαιώματα εδώ η αναφορά στις διμερείς συμφωνίες νομίζουμε πως δεν είναι απαραίτητη γιατί η αρχή είναι πως τα κράτη-μέλη δεν ξερούνται από τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την μη επιστροφή και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων άσχετα από οποιαδήποτε συμφωνία μπορεί να έχουν με τρίτες χώρες σε σχέση με αυτά τα θέματα. Και τέλος, η υποχρέωση αναφοράς, αυτό είναι ένα θέμα που θέλουμε να το σκεφτούμε περισσότερο, για να δούμε πώς θα μπορούσαμε καλύτερα να ανταποκριθούμε σε αυτή μας την υποχρέωση. Ευχαριστώ. Έχετε κάτι ακόμη να προσθέσετε κυρία Μάισνερ. Όχι, ευχαριστώ. Όχι, ευχαριστώ. Ας να συνεχίσει κάποιος άλλος. Να σας υπενθυμίσω ότι αύριο ψηφίζουμε για τη γνωμοδότηση αυτή. Θα σταματήσουμε μέχρι τις 4 ε, παρατέταρτο και θα περάσουμε στην έκθεση Μπαχ όταν έρθουν και οι σκιώδεις εισηγητές. Κάνουμε λοιπόν αυτή τη σύντομη διακοπή μέχρι τις 15.45 και ίσως οι συνεργάτες των πολιτικών ομάδων μπορούν να πάνε και να εντοπίσουν τους βουλευτές τους γιατί όπως βλέπετε εδώ πέρα μας έχει φάει η μοναξιά επειδή είμαστε εμείς και ο Κούκος. 15 λοιπόν. Okay, colleagues. Καλώς αγαπητοί συναδελφοί. Επαναρχίζουμε την συνεδρίαση και το επόμενο θέμα είναι η μεταρρύθμιση του κανονισμού για τα δικαιώματα των επιβατών με την παρουσίαση της έκθεσης από τον κύριο Μπαχ και μετά θα δώσω το λόγο στον κύριο Μάιερ εξ ονόματος της Επιτροπής ΙΜΚΟ για τους καταναλωτές και την εσωτερική αγορά και μετά θα δώσω το λόγο στους σκιώδεις. Μεταρρύθμιση λοιπόν των ε, του κανονισμού για τα δικαιώματα των επιβατών. Τζόρτζ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, να σας δώσω μερικές βασικές πληροφορίες σε σχέση με την έκθεσή μου που αφορά τη μεταρρύθμιση του κανονισμού για τους επιβάτες ε, αεροπορικών εταιριών για να υπάρξει μια πλήρης ε, παρουσίαση. Όπως αναφέρω και στην αιτιολογική σκέψη της έκθεσης, εγώ τονίζω την ανάγκη να υπάρξει μια ενίσχυση και μια εδραίωση των δικαιωμάτων των επιβατών. Η κατάσταση όπως έχει σήμερα δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική και δεν υπάρχει παρά μόνο ε, εμβαλωματική πολλές φορές εφαρμογή των κανονισμών σε σχέση με τους επιβάτες. Αν δούμε καλύτερα τώρα την πρόταση της Κομισιόν θα πρέπει να διαπιστώσουμε ότι σε σχέση με την τωρινή κατάσταση δεν μας προσφέρει καμιά ιδιαίτερη υποστημενή αξία σε ό,τι αφορά τους επιβάτες. Κάποια παραδείγματα. Υπάρχει μια αύξηση του χρόνου καθυστέρησης που δίδει δικαιώματα στους επιβάτες από 3 ώρες πηγαίνει στις 5 ώρες και για τις ε, πτήσεις μεγάλης διάρκειας μέχρι και, 12, μέχρι και 9 ή 12 ώρες. Επίσης, περιορισμούς του δικαιώματος στέγασης για έκτακτες περιπτώσεις σε 3 νύχτες επί 100 ευρώ και επίσης 12 ώρες για να μπορέσουν να μεταφέρουν οι επιχειρήσεις τους ε, επιβάτες με τα δικά τους μέσα προτού γίνει μια αναδιάταξη της, διαδρο... της διαδρομής και καμία αλλαγή σε ό,τι αφορά τους κανόνες για τις βαλίτσες, για τη διαφάνεια των τιμών ή για την αντιμετωπίση πτώχευσης των επιχειρήσεων. Για όλους αυτούς τους λόγους εγώ πάντα τονίζω την εξής αρχή, ότι οι επιβάτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν θα έχουν αυτόματα την εφαρμογή των δικαιωμάτων τους. Θα πρέπει οι επιβάτες να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και γι' αυτό να μπορούν να κάνουν τις διεκδικήσεις τους έναντι των μεγάλων επιχειρήσεων στον τομέα αυτό. Και εδώ πολλές φορές υπάρχει μια βεβαιότητα για τους επιβάτες, γιατί είναι πολύπλοκη η διαδικασία. Πολλοί, πολλοί επιβάτες λόγω του υψηλού κόστους και της, ε, του βάρους μιας διαδικασίας ενώπιον των δικαστηρίων δεν προβαίνουν σε συνέχιση αγωγών κατά των επιχειρήσεων για το γεγονός ότι δεν έχουν πάρει τις απαραίτητες υπηρεσίες. Αν συγκρίνουμε ορισμένα αριθμητικά στοιχεία, <clears throat> μόνο για περίπου 1% των πτήσεων που βρίσκονται στον τομέα εφαρμογή προκύπτουν προβλήματα για τα οποία υπάρχει διεκδίκηση των, των επιβατών. Μόνο περίπου 2% των επιβατών που έχουν το δικαίωμα σε αποσημείωση διεκδικούν αυτό το δικαίωμα για 100 πτήσεις με 100 επιβάτες κάθε μία σημαίνει μόνο 2 στους 10.000 επιβάτες. Και δεν είναι σίγουρο ότι τελικά αυτοί οι 2 στους 10.000 θα πάρουν την αποζημίωση. Επομένως αυτό δείχνει ότι κατά τη δική μου εκτίμηση η επιβάρηση των επιχειρήσεων ιδιαίτερα, των αεροπορικών επιχειρήσεων ιδιαίτερα χαμηλή. Με εντυπωσιάζει ιδιαίτερα μια δήλωση της Κομισιόν και παραθέτω. Το υψηλότερο κόστος θα οδηγήσει σε επιχειρήσεις ώστε να ελαχιστοποιήσουν το κόστος που συνδέεται με την εφαρμογή των κανόνων και επομένως να προσπαθήσουν να μειώσουν τα δικαιώματα των ε, επιβατών. Αυτό είναι μια παραδοχή ουσιαστικά ότι δεν σέβονται οι επιχειρήσεις, οι αεροπορικές εταιρείες τα δικαιώματα των επιβατών. Και εμείς θα πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια να, να εφαρμόσουμε τον νόμο όπως βολεύει τις εταιρείες. Αυτό δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Η νομολογία που υπάρχει για τα θέματα αυτά ε, έχει εδρεωθεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Υπήρξαν 39 διαδικασίες οι οποίες έχουν καταγραφεί για τα θέματα αυτά. Και θα αναφέρω μονάχα δύο τέτοιες περιπτώσεις, το λεγόμενη απόφαση Sturgeon του 2009, που αποφάσισε ότι οι επιβάτες όταν υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση έχουν το δικαίωμα για αποζημίωση. Και επίσης αυτό επιβεβαιώθηκε στην περίπτωση Nelson το 2012. Η πρόταση της Κομισιόν όμως έχει λάβει υπόψη αυτές τις ε, αποφάσεις και την ομολογία, αλλά τις έχει και αποδυναμώσει. Για την περίπτωση Sturgeon, ενώ ήταν το δικαίωμα, το δικαίωμα αποζημίωση ήδη σε τρεις ώρες, η Κομισιόν τα μεταφέρει αυτά σε πέντε, 9 ή 12 ώρες αντιστοίχως. Πιστεύω λοιπόν ότι από αυτά τα παραδείγματα μπορούμε να κατανοήσουμε τι μπορεί να συμβεί. Έχετε μια πτήση από το Λονδίνο στη Νέα Υόρκη που κανονικά φεύγει στις 3 ώρα το απόγευμα, έχει μια καθυστέρηση 11 ωρών. Και επομένως μόνο στις 2 ώρα το επόμενο πρωί έχει κανείς δικαίωμα κάποιας αποζημίωσης. Με τους κανονισμούς, αν φύγει το αεροπλάνο τότε, πιο πριν, δεν πρόκειται να πάρει καμία απολύτως αποζημίωση. Γι' αυτό τονίζω ότι πρέπει να επαναφερθεί το όριο των τριών ωρών για πτήσεις μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πέντε ωρών για πτήσεις μακράς αποστάσεως. Η ενοποίηση των ε, χρόνων αποζημίωσης και των ποσών που έχουν να κάνουν με την αποζημίωση για πτήσεις μέχρι 3.500 χιλιόμετρα στα 300 ευρώ και 600 ευρώ για πτήσεις που είναι μεγαλύτερης αποστάσεως Αυτά θα οδηγούν σε μεγαλύτερη σαφήνεια και καλύτερη ε, κατανόηση των καταναλωτών. Ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι η λεγόμενη ε, απόφαση Βαλεντίν Χέρμαν από το 2008 που κάνει σαφές ότι τα τεχνικά προβλήματα δεν θεωρούνται αφεαυτών έκτακτες περιστάσεις. Στην έκθεσή μου τονίζω εγώ ότι τα τεχνικά προβλήματα είναι μια φυσιολογική δυσκολία και πρόκληση που περιλαμβάνεται στη λειτουργία μια αεροπορική επιχείρηση και μόνο σε ορισμένε περιπτώσει, όταν υπάρχει ανωτέρα βία λόγω φυσικών καταστροφών ή σαμποτά, μπορούν να θεωρηθεί ότι δίνουν ελαβή σε έκτακτε καταστάσει. Δεύτερον, έχουμε το γεγονό ότι οι επιβάτε δεν γνωρίζουν ποια είναι τα δικαιώματά του και γι' αυτό το λόγο εγώ τόνισα ότι πρέπει να υπάρξει το δικαίωμα πληροφόρηση, το οποίο πρέπει να ενισχυθεί και να υπάρχει πάντα σαφής παρουσία συνομιλητών από τις ε, αεροπορικές επιχειρήσεις στα αεροδρόμια, ώστε να αντιμετωπίσουν και να δώσουν συγκεκριμένες πληροφορίες και βοήθεια στους επιβάτες όταν αυτό απαιτείται. Ένα άλλο πολύ σημαντικό πακέτο είναι και η διαφάνεια των τιμών. Και εδώ είναι απαραίτητο να υπάρχει μέσα στις γενικές συνθήκες όταν κανείς κλείνει ένα εισιτήριο να υπάρξει μια μεγαλύτερη σαφήνεια ώστε να μην υπάρχουν αμφισημίες όταν κανείς κλείνει ένα εισιτήριο και να ξέρουν οι επιβάτες ποια είναι τα δικαιώματά τους. Με τον τρόπο αυτό θα αποφεύγεται ορισμένε εταιρείε να ζητούν πρόσθετα τέλη για το κλείσιμο ενό εισιτηρίου και να έχουν τέτοια τέλη τα οποία πολλέ φορέ ξεπερνούν και την τιμή του εισιτηρίου ή να ζητούν πρόσθετα ποσά για να μπορεί κανεί να μεταφέρει μία βαλίτσα ή μία ομπρέλα ή οτιδήποτε άλλο. Επίσης, ό,τι αφορά την πτώχευση των αεροπορικών εταιριών, εγώ υπενθυμίζω την αίτηση του Κοινοβουλίου από προηγούμενα ψηφίσματα. Πρέπει οι επιβάτες για περιπτώσεις πτώχευσης των εταιριών να είναι ε, εξασφαλισμένοι, να είναι ασφαλισμένοι, όπως αναφέρει και η οδηγία για τα ε, επιμέρους ταξίδια. Η πρότασή μου είναι ότι αυτό μπορεί να γίνει μέσα από ένα ταμείο το οποίο θα δημιουργήσουν οι ίδιες εταιρείε. Σε ό,τι αφορά τις καθυστερήσεις στην πίστα των αεροπλάνων. Πιστεύω ότι όπως η Κομισιόν έχει προτείνει, πέντε χρόνια χρόνος αναμονής είναι υπερβολικός και προτείνω ότι μετά από δύο ώρες οι επιβάτες θα έχουν το δικαίωμα να εγκαταλείψουν το αεροσκάφος το οποίο δεν έχει ακόμα απογειωθεί. Και να τονίσω ότι προσπαθώ να επιτύχω μια ισορροπία σε όλα αυτά τα θέματα, τονίζω ότι υπάρχουν και ορισμένε άλλες προτάσεις οι οποίες ε, αναφέρονται και στι ανάγκε των αεροπορικών εταιριών. Για την πολιτική όταν κανεί δεν εμφανίζεται, τονίζω ότι οι αεροπορικέ εταιρείε δεν μπορούν να αρνηθούν το ταξίδι επιστροφή αν ο επιβάτη δεν έχει κάνει το ταξίδι αλέ. Θα ήθελα λοιπόν να υπάρχει και μια αντίστοιχη αντιμετώπιση για ένα ταξίδι το οποίο έχει διάφορα τμήματα διαδρομών. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η ε, ανταποκρίσεις που χάνονται από τον επιβάτη. Καταρχήν θα πρέπει να υπάρχει η ευθύνη στην πρώτη εταιρεία η οποία έχει προκαλέσει την καθυστέρηση. Νομίζω ότι εδώ και για μικρές καθυστερήσεις μπορεί να προκύψει δικαίωμα αποζημίωσης του επιβάτη. Όταν όμως έχει ξεπεράσει τα 90 λεπτά καθυστέρηση και έρχεται ο επιβάτη με καθυστέρηση πάνω από 3 ώρε ή πέντε ώρε. Τότε θα πρέπει να μπορεί να έχει το δικαίωμα ε, αποζημίωση λόγω αυτή τη αρχική καρτιστέ. Ένα άλλο στοιχείο είναι η 5 ωρε τοτε θα πρεπει να μπορει να εχει το δικαιωμα αποζημιωση λογω αυτη τη αρχικη καθυστερησης ενα αλλο στοιχειο ειναι η εφαρμογη και η αστυνόμευση. Εδώ έχω προτείνει μεταξύ άλλων να ακολουθήσουμε αυτά που λέει η οδηγία για την Alternative Dispute Resolution, την εναλλακτική επίλυση διαφορών, που υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να έχουν εθνικούς φορείς για την διαιτησία και την επίλυση την εξοδικαστική διαφορών χωρίς να είναι υποχρεωμένοι οι επιβάτες να προσφεύγουν πάντα στα δικαστήρια. Για την προετοιμασία αυτής της έκθεσης εγώ έχω ερθισόμενους και ε, ενεργούς στον τομέα αυτό και έχω ακούσει τα επιχειρήματά τους. Απλώς πρέπει να πω ότι με έχει ενοχλήσει η κάπως αρνητική στάση ορισμένων εκπροσώπων του αεροπορικού κλάδου που δίνουν την εντύπωση ορισμένε φορές ότι ο επιβάτης για αυτούς είναι ένα εμπόδιο σε ό,τι αφορά την παραγωγή επιβατοχιλιόμετρων. Πιστεύω ότι αυτό είναι πραγματικά πάρα πολύ ανησυχητικό, γιατί πάντα εγώ θεωρώ ότι πρέπει κανείς να νιώθει ως επιβάτης ότι είναι ένα είδος καλεσμένου στο αεροπλάνο που έχει δικαιώματα τα οποία γίνονται σεβαστά. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω την αντίδραση των συναδέλφων και είμαι σίγουρο ότι τι επόμενε εβδομάδε θα μπορέσουμε να έχουμε μια πλήρη και εντατική συζήτηση για τα διάφορα πολιτικά σημεία που έχουν να κάνουν αυτή την πρόταση. Σα ευχαριστώ για την προσοχή σα. Ευχαριστούμε κύριε Μπάκ. Ο κύριο από την ΕΜΚΟ. Ευχαριστώ. Η έκθεσή μου στην ΙΜΚΟ είναι στη μετάφραση αυτή τη στιγμή. Σύντομα θα είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες. Αλλά από αυτά που ακούσαμε πιστεύω ότι υπάρχει μια μεγάλη σύμπνοια μεταξύ ημών και του κυρίου Μπαχ. Η ΙΜΚΟ είναι αρμόδια για την προστασία των καταλατών και γι' αυτό η εστίασή μου βρίσκεται στα δικαιώματα των καταναλωτών και το δίκαιο των καταναλωτών που βέβαια θα πρέπει να συμβαδίζει με τα θεμητά συμφέροντα των αεροπορικών εταιρεών. Αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι, όπως είπε και ο κύριος Μπαχ, να είναι πιο συνεκτική η διαδικασία αποζημίωσης με τα χρονικά όρια και με δύο ποσά ανάλογα με την περίπτωση. Επίσης, θα πρέπει στην τιμή του εισιτηρίου να απελαμβάνονται όλα τα τέλη. Δεν μπορεί κανείς να πληρώνει 29 ευρώ για μία πτήση. Δεν μπορεί στη συνέχεια να του επιβάλλονται τέλη τα οποία ξεπερνούν την τιμή του εισιτηρίου. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να περιορίζονται τα πρόσθετα τέλη στο εισιτήριο. Σε ό,τι αφορά την αποζημίωση για τις ζημίες, πιστεύω ότι εδώ ακόμα είναι κάπως ασαφής η διατύπωση. Θα πρέπει να είμαστε σαφέστεροι και να πούμε ότι όταν υπάρχουν δυνατότητες περαιτέρω ζημίας, δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι έχει κλείσει το θέμα αυτό. Πάντα Μπορεί κανείς να ζητήσει περισσότερα σε δικαστικό επίπεδο και έχει το δικαίωμα να το κάνει αυτό. Δεν σημαίνει ότι χάνει κάθε δικαίωμα ε, διεκδίκησης. Επίσης για την καθυστέρηση της στην πίστα, συμφωνώ με τον κύριο Μπαχ, για τις ε, πρόσθετες ε, ε, για τις περιπτώσεις όταν υπάρχει μια καθυστέρηση η οποία δεν οφείλεται στην αεροπορική εταιρεία, επίσης συμφωνώ. Έχω και μερικά ακόμα πρόσθετα στοιχεία το θέμα της παραγραφής παραδείγματος χάρη, αυτό είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με το εθνικό δίκαιο, αλλά επειδή εδώ έχουμε ένα ε, ευρωπαϊκό νομοθέτημα, θα πρέπει να έχουμε ένα διάστημα δύο ετών τουλάχιστον το οποίο να ισχύει για όλες τις περιπτώσεις, ώστε να μην υπάρχει κάποια ασάφεια σε ό,τι αφορά την επιβροφή για τα θέματα αυτά. Το θέμα των έκτακτων περιστάσεων βέβαια είναι ένα σταυρόλεξο για όλους και ένα πονοκέφαλος. Είναι πολύ δύσκολο να ξέρουμε πότε μπορεί αυτό να είναι σαφές. Εγώ νομίζω ότι η Κομισιόν δεν το έχει παρουσιάσει πολύ σωστά. Όπως είπε και ο κύριος Μπαχ, θα πρέπει να υπάρχει μεγάλη σαφήνεια για τα τεχνικά προβλήματα. Μόνο λοιπόν τα τεχνικά προβλήματα πέραν αυτών τα οποία μπορεί να περιμένει κανείς από ένα έλεγχο των αεροσκαφών μπορούν τέτοια <clears throat> προβλήματα να θεωρηθούν προβλήματα για τα οποία δεν είναι υπεύθυνη η αεροπορική εταιρεία. Όλα αυτά τα οποία υπόκειται στην κανονική συντήρηση ενός αεροσκάφους και στον έλεγχο του αεροσκάφους είναι υπόθεση της ε, αεροπορικής εταιρεία και άμα δεν γίνει σωστή συντήρηση δεν φταίει ο επιβάτης. Επίσης, <clears throat> οι καθυστερήσει ή τα προβλήματα λόγω των καιρικών συνδικών. Αυτό είναι ένα δύσκολο πρόβλημα. Και εγώ πέρασα σε μία περίπτωση όπου μου είπαν ότι ήταν κακές οι καιρικέ συνθήκε, ενώ στην πραγματικότητα δεν ήταν οι καιρικέ συνθήκε οι οποίε οδήγησαν στο πρόβλημα. Υπήρχε συμφόρηση και λόγω αυτής της συμφόρησης έπρεπε να καθυστερήσει η απογείωση των αεροσκαφών και αυτό οδήγησε σε μια καθυστέρηση. Αυτό όμως είναι επιχειρηματικές αποφάσεις και όχι αποφάσεις οι οποίες έλκονται από τις κεντρικές συνθήκες και πρέπει να είμαστε σαφείς εδώ. Το δικαίωμα σε πληροφόρηση και δυνατότητα υποβολής παραπώνων. Εδώ δεν υπάρχει μέχρι στιγμής πραγματικό δικαίωμα διεκδίκησης από τους πολίτες. Θα ήθελα να υπάρχει μια πραγματική προστασία που να εξασφαλίζει ότι μπορεί να υποβάλει παράπονα χωρίς να υπόκειται σε κυρώσεις. Είναι σημαντικό λοιπόν να μπορεί ο πελάτης να έχει μία ε, απάντηση και να του δίδονται και τα έγγραφα τα οποία είναι απαραίτητα για να ελέγξει κατά πόσο γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Θα πρέπει να είναι απαραίτητο λοιπόν να μην χρειάζεται κανείς να πάει στα δικαστήρια για να διεκδικήσει τα έγγραφα τα οποία εδραιώνουν τα δικαιώματά του. Ο επιβάτης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να έχει στα χέρια του όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται για να μπορεί ο ίδιος να αποφασίζει αν μπορεί να ευδοκιμήσει η αίτηση του στο δικαστήριο πριν πάει στο δικαστήριο. <clears throat> Γενικά λοιπόν, όπως είπε και ο κύριος Μπαχ, οι επιχειρήσεις προσπαθούν όταν υπάρχουν παράπονα των ε, επιβατών να αποφύγουν την εφαρμογή δικαιωμάτων τα οποία είναι δεδομένα. Αυτό είναι παραγνώριση του ευρωπαϊκού δικαίου και παραβίασή του. Επομένως, εδώ πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να έχουμε μια καλύτερη αντιμετώπιση και να υπάρχει δυνατότητα επιβολής κυρώσεως. Το θέμα του νομίσματος στο οποίο γίνεται η αποζημίωση, αυτό μπορεί να φαίνεται τετριμένο θέμα, αλλά πιστεύω ότι στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να το αναφέρουμε με στρογγυλούς αριθμούς σε ευρώ, οπότε να έχουμε κάποιο ποσό το οποίο θα είναι εύληπτο. Σας ευχαριστώ εν τέλει για την ευκαιρία να έρθω ενώπιον της Επιτροπής σας και να λάβω το λόγο. Ενώπιον σας έχουμε μεγάλη σύμπνοια και συμφωνία με τον εισηγητή, απλώς με ορισμένα θέματα τα οποία ανέφερα προηγουμένως, τα οποία θα είναι χρήσιμο να τα διαλευκάνουμε περισσότερο και έτσι με τον τρόπο αυτό να καταλήξουμε σε μια σωστή πρόταση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Και τώρα, εξ το των ομάδων, η κυρία Βανό για τους Σοσιαλιστέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα εν γέννη να χαιρετήσω την πολύ καλή δουλειά που έκανε ο συνάδελφος Μπακ και να τον ευχαριστήσω γιατί αποπειράθηκε να λάβει υπόψη και να βελτιώσει τα διάφορα σημεία της πρότασης ε, που έπρεπε να βελτιωθούν και αυτό πάντοτε μέσα στο πλαίσιο της υπεράσπισης των ε, επιβατών έχοντας υπόψη του να διευκρινίσει όσο γίνεται τα πράγματα και να απλοποιήσει γιατί η ε, νομική ασφάλεια είναι πολύ ουσιώδης εδώ για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. τώρα Βέβαια θα πρέπει να μιλήσω γενικά για ολόκληρη την έκθεση. Είμαι θετική απέναντι στις διατάξεις που είναι πιο ευνοϊκές προς τους καταναλωτές και τους, και τους επιβάτες. Η ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στους ε, ανάπηρους στα άτομα με περιορισμένη κινητικότητα. Στον καθορισμό της άρνησης επιβίβασης, ε, στην ενίσχυση της προστασίας των επιβατών σε περίπτωση πτώχευσης μιας εταιρείας, την υποχρέωση κάθε εταιρεία να έχει ένα άτομο επαφή σε όλα τα αεροδρόμια Όλα αυτά είναι θετικά. Σε πιο συγκεκριμένα σημεία, ιδιαίτερα όσον αφορά τις διάφορες προθεσμίες, έχω την εντύπωση πως και εκεί θα μπορέσουμε να βρούμε μια συμφωνία, ακόμα και αν μπορούμε ακόμα να συζητήσουμε τις ε, διαδικασίες. Ο νέος υπολογισμός των καθυστερήσεων, ε, καθώς και η κατάργηση της προθεσμίας των δύο ωρών πριν από την ε, ανάληψη ευθύνη είναι ενδιαφέρουσες, ακόμα και αν υπάρχουν διαφορές 10, 15, 30 λεπτά ε, ίσως κάτι τέτοιο δεν χρειάζεται να οδηγεί σε άμεση παροχή αναψυκτικών. Ένα από τα σημεία όμως που μπορεί να προκαλέσει μεγάλη συζήτηση, ιδιαίτερα από πλευρά των ε, αεροπορικών εταιριών, είναι φυσικά το, τα κατόφλια μετά τα οποία 5, 9, 12 ώρες δηλαδή, που μειώνονται στις 3 και 5 ώρες όσον αφορά τις αναμονές. Για, ίσως θα μπορούσαμε να συζητήσουμε να καταργήσουμε την το τελευταίο κομμάτι πτήσεων άνω των 6.000 χιλιόμετρων, ωστόσο συμμερίζομαι τη γνώμη του εισηγητή ότι 5 ώρε για ενδοευρωπαϊκέ πτήσει είναι υπερβολικό. Σε περίπτωση των αποζημιώσεων, διευκρινίζω τη βούλησή μα να ε, συνηθούν ε, θελοντικέ συμφωνίε, γιατί κάτι τέτοιο είναι πιο ενδιαφέρον για ε, τον ε, επιβάτη παρά η αποζημίωση. Όσον αφορά τώρα τις, τις ε, ανταποκρίσει, συμφωνώ ότι θα πρέπει να μεταφέρεται η ευθύνη στην εταιρεία που είναι υπεύθυνη για την καθυστέρηση. Όσον αφορά όμω την αποζημίωση, νομίζω πω ε, πρέπει να συζητήσουμε τι διαδικασίε τόσο όσον αφορά τα ποσά, όσον αφορά και τη διάρκεια τη αρχική ε, καθυστερήση, ακόμα και αν η προσέγγισή σα είναι ενδιαφέρουσα. Θα μπορούσαμε επίση να σκεφτούμε, και αυτό νομίζω είναι σημαντικό, μια καλύτερη ενημέρωση όσον αφορά του επιβάτε για τη διάρκεια τη ανταπόκριση και τον κίνδυνο αναμονή στο τράνζιτ για πολύ λίγο χρόνο από τη στιγμή της κλίση, του κλεισίματος των εισιτηρίων. Ε, επίσης νομίζω πως μπορούμε να διατηρήσουμε διατάξεις ε, για να μην υπάρξει καταχρηστική ε, χρέωση από πλευράς των εταιριών που αναλαμβάνουν τους επιβάτες σε last minute. Τώρα, άμεση ανάληψη του ε, επιβάτη από την εταιρεία και αυτή η πρότασή σας είναι ενδιαφέρουσα. Είμαι υπέρ δε του περάσματος από το, στο 1,5 εκατομμύριο επιβατών για να φτιαχτούν σχέδια διαχείρισης επίγουσας κατάστασης και πρέπει να προχωρήσουμε περισσότερο για τη διευκρίνηση του ρόλου του καθενός. Αερολιμένες, εταιρείε, δημόσια αρχή, ανάλογα με την περίσταση. Ένα άλλο ευαίσθητο σημείο, δηλαδή άρνηση ε, επιβίβασης για τους ε, όσο αυτούς που δεν εμφανίζονται δηλαδή, θα πρέπει να το διευκρινίσουμε και ίσως να φτιάξουμε και ένα σύστημα στις εταιρείες που θα μπορούν να πουλήσουν τη θέση αφού ε, θα είναι βέβαιοι ότι ο επιβάτης δεν είχε σκοπό να χρησιμοποιήσει το δεύτερο τμήμα του ταξιδιού, το ίδιο και στις πτήσεις ανταπόκρισης και όχι μόνο στα Λερετούρ. Πάντως κανείς δεν θα ήθελε να δει να συνεχίζεται αυτή η πολιτική μονομερούς ακύρωσης για το θέμα των αποσκευών. Και εδώ συμμερίζομαι τη θέση του εισηγητή όσον αφορά τις ε, τσάντες duty free και τις ε, τσάντες χειρός καθώς και τα όργανα μουσικής. Ωστόσο θα μπορούσαμε να μείνουμε στην μία αποσκευή καταγεγραμμένη στο πλαίσιο της ε, διαφάνειας των τιμών που είναι επίσης ένα θετικό στοιχείο της έκθεσης. Πάντα σε θέματα διαφάνειας και ενημέρωσης να χαιρετήσω τη βούληση για, την σύνταξη ενός εντύπου δήλωσης με συγκεκριμένα δικαιώματα καθώς και τη γλώσσα και το τι τύπο που θα πρέπει να χρησιμοποιείται και πρέπει αυτό να το συζητήσουμε, είναι πολύ σημαντικό. Επίσης είναι σημαντικό να διευκρινιστούν οι ευθύνε όσον αφορά την ε, ε, ε, αναγραφή των προσωπικών στοιχείων. Ε, θα πρέπει ο επιβάτης να γνωρίζει ποιες είναι οι πρακτικές συνέπειες, αν αρνηθεί ή ξεχάσει να δώσει τις πληροφορίες αυτές. Τώρα, όσον αφορά τις έκτακτες περιστάσεις, ο εισηγητής θέλησε να λάβει υπόψη πιο συγκεκριμένα το, την απόφαση Βαλαντά. Είναι σημαντικό όμως να προσθέσουμε και ένα θετικό κατάλογο περιστάσεων, ένα κατάλογο όπου έχουν αρχίσει να εργάζονται οι αντίστοιχες ομάδες και πιστεύω πως ε, οι έκτακτες περιστάσεις είναι περιστάσεις που από τη φύση τους ή λόγω της προέλευσής τους ξεφεύγουν από τον έλεγχο του, της αεροπορικής εταιρείας και δεν θα μπορούσε να τις έχει αποφύγει ακόμα και αν είχε λάβει όλα τα λογικά μέτρα. Όσον αφορά τα τους ONA, πιστεύω ότι ναι, θα πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος τους ε, ελέγχου και αποτροπής, αλλά να υπάρξει και εναρμόνιση ανάμεσα στα κράτη. Γιατί κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο όσον αφορά την, τον ενιαίο χαρακτήρα του νόμου. Ε, πιστεύω λοιπόν πως θα μπορέσουμε να βρούμε καλές λύσεις. Ευχαριστώ και πάλι τον εισηγητή για την εργασία του και ως σκιώδης στην Επιτροπή Μεταφορών αλλά και Αντιπρόεδρο τη ΣΥΜΚΟ που ασχολείται με τα δικαιώματα του καταναλωτή, είμαι πεπισμένη πω μπορούμε να βρούμε ισορροπία. Διότι οι επιβάτε που εξυπηρετούνται καλύτερα, όπως, ε, σαν να είναι προσκεκλημένοι, με όλη την απαραίτητη προσοχή, επειδή ακριβώς θα δουν πως η ασφάλειά τους αυξάνεται θα έχουν περισσότερη εμπιστοσύνη στις αεροπορικές εταιρείες και άρα θα συμβάλλουν επίσης στο να αυξηθεί και να ενδυναμωθεί η καλή εικόνα αυτών των εταιρείων και άρα κατά συνέπεια θα συμβάλλουν στην ανάπτυξή τους σε ένα πλαίσιο ανταγωνιστικό πιο δίκαιο και πιο ρυθμιζόμενο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει. κυρία Μάισνερ. Έχω ήδη αναφέρει στον εισηγητή, στον πρόεδρο, υπήρξαν πολλοί οι οποίοι έχουν διαμαρτυρηθεί για την έλλειψη πληροφοριών από το αεροδρόμιο των Βρυξελών. Αυτό δεν είναι ιστορία με τις αεροπορικές εταιρείε. Είναι προβλήματα που έχουν να κάνουν με το αεροδρόμιο. Πολλές φορές χρειάστηκε να περιμένουμε μισή ώρα στα διαβατήρια ή υπήρξαν ε, κάποια, κάποια γκρουπ τα οποία έχουν ταλαιπωρηθεί για καθυστερήσει και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το προσθέσουμε λοιπόν σε όλα αυτά τα πράγματα. Α, εγώ συνεχίζω στα αγγλικά γιατί στα αγγλικά μου έχουν δώσει το κείμενο που θα διαβάσω. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την πολύ καλή εργασία του. Η συνεργασία ήταν ιδιαίτερα καρποφόρα και μπορούμε να δούμε και από το σχέδιο του εισηγητή ότι έχουν περιληφθεί πολλά σημεία τα οποία έτυχαν συζήτηση και κάποια σημεία τα οποία θέλω να τονίσω. Εγώ υποστηρίζω ότι πέντε ώρες καθυστέρηση είναι πάρα πολύ μεγάλο διάστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου οι περισσότερε πτήσει είναι γύρω στι δύο ώρε. Και στην περίπτωση Sturgeon, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θεώρησε ότι ήδη τρει ώρε είναι μεγάλη καθυστέρηση. Δεύτερον, υποστηρίζω την ε, ε, αλλαγή λόγω σφαλμάτων που είναι δωρεάν και την ε, δυνατότητα να ε, μην ακυρώνται πτήσεις για να προστατεύσουμε τις περιφερειακές ε, εταιρείες η αλλαγή σε σχέση, η καθυστέρηση σε σχέση με την ασφάλεια θα πρέπει να μην οδηγήσουν σε προβλήματα ασφαλείας για τους ε, ε επιβάτες. 300 ευρώ λοιπόν θα πρέπει να είναι το κατώτατο όριο. Θα πρέπει το ποσό να εξαρτάται από την τιμή του εισιτηρίου. Κάτι ακόμα το οποίο πρέπει να αναφέρουμε είναι οι σωρευτικές καθυστερήσεις λόγω έκτακτων περιστώσεων. Σε πόσες περιπτώσεις θα πρέπει να ισχύει αυτό, πόσες πτήσεις θα πρέπει να καλύπτει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τις μικρές εταιρείες που δεν έχουν πολλά αεροσκάφη στη διάθεσή τους. Κάτι ακόμα που χρειάζεται διευκρίνηση είναι το θέμα περιορισμών όταν που υπάρχουν μονάχα δύο πτήσεις την εβδομάδα ή κάτι τέτοιο, πολύ λίγες πτήσεις. Κάτι ακόμα που πρέπει να καθοριστεί είναι οι πρόσθετε αποσκευέ. Εγώ υποστηρίζω ότι ο επιβάτη θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να φέρει κάποια προσωπικά στοιχεία ή όνια από το αεροδρόμιο επιπλέον, αλλά δεν μπορεί να είναι απεριόριστο το ποσό ή το μέγεθό του. Νομίζω ότι έχει κάνει πολύ καλή δουλειά ο εισηγητή και έχει δημιουργήσει μια πολύ καλή βάση διαπραγματεύσεων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Μάικλ, για του πράσινου. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή και τους δύο εισηγητές, αναφέρομαι και στον εισηγητή της ΣΥΜΚΟ, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι σήμερα ήρθε στην ώρα του το αεροπλάνο μου. Ήρθα στην ώρα μου. Τι έγινε μετά όμως, περίμενα μισή ώρα τη βαλίτσα μου. Και αυτό γίνεται πάντα. Άλλες φορές δεν έχετε στην ώρα το αεροπλάνο, τώρα ήρθε αλλά δεν ήρθε η βαλίτσα. Θα ήθελα να ξέρω η Κομισιόν μήπως έχει σκεφτεί να λάβει και αυτά τα θέματα. Γιατί υπάρχει μόνιμα μια παραβίαση των δικαιωμάτων των επιβατών. Λέει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο πέντε ώρες. Κάνω μια συμφωνία με την εταιρεία, κάνω μια σύμβαση με την εταιρεία και την πληρώνω εγώ την ύφη. Εγώ θεωρείται ότι είμαι ο φταίχτης γιατί η εταιρεία δεν έχει προσφέρει τις υπηρεσίες. Και έχουν κάποια, ε, κάποια δρομολόγια τα οποία δεν μπορούν να λειτουργήσουν αν κάποιος πρέπει να αλλάξει αεροπλάνο. Δεν μπορεί λοιπόν τα, να γίνονται αυτά τα δρομολόγια τα οποία δεν μπορούν να τηρηθούν. Θα πρέπει να μην επιτρέπεται σε εταιρείε να έχουν τέτοια δρομολόγια και τέτοιες ανταποκρίσεις και δεν θα πρέπει να το πληρώνουν αυτό οι επιβάτες. Εάν ήταν τελικά στην ώρα της όλα τα αεροπλάνα, τότε δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα αποζημίωση. Αυτό θα πρέπει να μπει στο μυαλό των αεροπορικών εταιριών και όχι να κάνουν κόλπα για να μην αποζημιώνουν τους επιβάτες. Το 70% όλων των επιβατών δεν έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τις αποζημιώσεις που ε, δικαιούνται. Αποφασίσαμε όλοι στις 5 ώρες να υπάρχει αποζημίωση. Αυτό λέει και η Κομισιό και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο όχι λέει αυτό είναι πάρα πολύ, αυτό είναι και ένα χαστούκι και για την Κομισιό. Δεν μπορεί να λέει τώρα η Κομισιόν ότι δεν μας ενδιαφέρει η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και συνεχίζουμε σαν να μην γίνεται τίποτα. Άμα θέλω να πετάξω από τη Φραγκφούρτη στο Λος Άντζελες και έρχομαι μετά από 11 ώρες και 55 λεπτά καθυστέρηση, τι μου λέτε, δεν έγινε τίποτα γιατί δεν περάσετε τις 12 ώρες. Δεν καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό να έχει καθυστερήσει κανείς τόσο πολύ. Πρέπει να αλλάξει ξενοδοχείο, δεν έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει το δρομολόγιο του. Λοιπόν, πού θα μείνω εγώ το βράδυ και πώς θα συνεχίσω την, ε, το ταξίδι μου. Δεν γίνεται αυτό και για τις έκτακτες περιστάσεις. Αυτό το παρουσιάζουν οι αεροπορικές εταιρείες σαν να γίνεται κάθε, δύο, και, και τρεις μέρες. Όταν το αεροπλάνο δεν είναι εν κινήσει και συμβεί κάτι, εντάξει τότε αυτό μπορεί να οφείλεται σε εξωτερικές συνθήκες. Όταν όμως το αεροπλάνο είναι ε, εν κινήσει τότε δεν υπάρχει καμία απολύτως αποζημίωση. Σκεφτείτε λοιπόν και ποια είναι η πίεση στους, πάνω στους πιλότες, πιλότους συγγνώμη, που υποχρεώνται πολλές φορές παρά το γεγονός ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο αεροπλάνο να πετάξουν για να μην δώσει αποζημίωση ε, η αεροπορική εταιρεία στους επιβάτες. Πώς μπορούμε λοιπόν να έχουμε τέτοιες ε, ε, ρυθμίσεις. Και δεν υπάρχει και μία ανεξάρτητη διαιτησία για τους, τις συνδρομικές μεταφορές. Τα καταφέραμε και δουλεύουν μια χαρά. Γιατί δεν μπορούμε να το έχουμε το ίδιο πράγμα για τις αεροπορικές πτήσεις. Να έχει κάποιος ένα τηλέφωνο που να του λέει πληροφορίες για αυτά τα οποία χρειάζονται. Και γι' αυτό αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι τα 90% αυτών που έχουν δικαίωμα σε αποζημίωση ξέρουν ότι είναι χρονοβόρα και βαριά η διαδικασία, δεν κάνουν απολύτω τίποτα. Και πρέπει να υπάρχει φυσικά και ένα δικαίωμα να μην περιορίζονται αυτόματα, να διατηρείται το δικαίωμα. Νομίζω οι εταιρείε αυτή τη στιγμή παίρνουν λεφτά από του Ευρωπαίου ε, φορολογούμενους. Έχουν επιδότηση για την κυροζήνη που χρησιμοποιούν στις εξωτερικές μεταφορές τους και αυτό ουσιαστικά ε, είναι επιδότηση του Ευρωπαίου πολίτη. Εμείς έχουμε δώσει 30 δισεκατομμύρια με την επιδότηση στην κυροζήνη σε αεροπορικέ εταιρείε και οι εταιρείε τραβάνε τα μαλλιά του και σχίζουν τα ημάτια του ότι δεν έχουν καθόλου λεφτά. Λοιπόν, αυτά τα οποία κάνουμε στου σιδηροδρόμου θα πρέπει να τα κάνουμε και ε, στι αεροπορικέ εταιρείε. Μετά από μία ώρα καθυστέρηση στα τρένα 25% του εισιτήριου πιβάτης μετά από τρεις ώρες το 50%. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να ισχύσει και στις ε, αεροπορικές εταιρείες. Και αν έχω πληρώσει 5.000 εισιτήριο πρώτης θέσης, τότε θα πρέπει να είναι ακόμα περισσότερο. Αυτή είναι λοιπόν η κατεύθυνση την οποία εγώ υποστηρίζω, να υπάρξει μια δυνατότητα αυτόματης διατησίας. Αν θέλουμε και για τις βαλίτσες, εάν θέλουμε να έχουμε λοιπόν μια ρύθμιση ενιαία ανταγωνισμού. Ό,τι ισχύει για το τρένο πρέπει να ισχύει και για το αεροπλάνο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ τον κύριο Πάκ και ζητώ συγγνώμη που δεν ήμουν εδώ. Άργησε η πτήση μου και κατέθεσα για το ε, παρέμπονο μου στην Κομισιόν. Έχασα κάποιες αρχικές παρατηρήσεις, ε, αλλά θέλω να σας ευχαριστήσω για το όσα κάνατε μέχρι στιγμής. Να ξεκινήσω λέγοντας πως βέβαια είμαστε σε κάποια... Θε... Ε, συμφωνούμε μάλλον γενικά, αλλά σίγουρα έχουμε θέμα ως Ηνωμένο Βασίλειο με το Γιβραλτάρ. Και μέχρι ότου λυθεί αυτό το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα κάνει καμιά αλλαγή, γιατί δεν θα μπορεί. Οπότε θέλω αυτό να το αναφέρω, είναι κάπως ευρύτερο από όλη την έκθεση. Και τώρα μπαίνω σε λεπτομέρειες. Ίσως ε, βεβαίως θα πρέπει όντως μετά από όλες αυτές τις υποθέσεις και με εκείνη την ε, στάχτη, την ηφαιστιακή που έγινε χαμός τότε, ε, φάνηκε πως έπρεπε να βρεθούν λύσεις. Είτε είναι οι αεροπορικές εταιρείε είτε είναι οποιοδήποτε, πρέπει να βρεθεί τρόπος να προχωρήσουμε. Και εφόσον δει κανεί την πρόταση της Κομισιόν, σίγουρα κατά τη γνώμη μας υπάρχουν πολύ θετικά στοιχεία. Όχι όλα, αλλά κάποια είναι θετικά. Και από τις 3 στις 5 ώρες να μετακινηθούμε πιστεύουμε ότι είναι καλή ιδέα. Γιατί είναι λιγότερο πιθανό να κυρώσει κανείς την πτήση από ότι με τις 3 ώρες. Πολύ σημαντική πρόταση αυτή λοιπόν και εδώ λοιπόν με τον κύριο Μπακ έχουμε διαφορετική θέση, θέλουμε να μείνουμε στο status quo. Τώρα, σε σχέση με τις έκτακτες περιστάσεις, πρέπει να, να προσέξουμε, ε, να δούμε πώς θα καθορίσουμε εκ νέου αυτό στις έκτακτες περιστάσεις. Υπάρχει ένας κατάλογος, έχει γίνει πολλή δουλειά γι' αυτό και εμείς ε, θα συμφωνήσουμε με τα όσα συμφωνούν όλοι για μια συμπεφωνημένη λίστα Δηλαδή το Συμβούλιο, η Κομισιόν και οι αεροπορικέ εταιρείε, γιατί είναι πολύ δύσκολο. Είναι δύσκολο να μιλάμε για έκτακτε συνθήκε, αλλά είναι πολύ δύσκολο όταν πρόκειται για τεχνικά ζητήματα. Εγώ θεωρώ κάποια πράγματα ότι είναι έξτρα, έκτακτα, αλλά όχι. Πάντως πρέπει να διευκρινιστούν. Ε, τώρα σε σχέση με την πρόταση της Κομισιόν για τις ανταποκρίσεις ε, δεν υπάρχει αρκετή κατανόηση. Αν σε καθυστερήσει κάποιος ε, και αν δεν είναι μόνο μια καθυστέρηση μιας μέρας, ε, μπορεί να υπάρξουν 24 ώρες καθυστέρηση λόγω κακου, κακοκαιρίας. Ποιος θα πληρώσει, ποιος θα αποζημιώσει, πώς λειτουργούν όλα αυτά. Ας πούμε, αν υπάρχουν τώρα δυσκολίε και είναι σωρευτικά και κρατήσει τρει μέρες, δεν μπορεί να δει κανεί δηλαδή μόνο την προηγούμενη πτήση. Πρέπει πολύ να προσέξουμε. Και κάτι πολύ καλό που είπε η κυρία Μάλιστερ είναι ότι πρέπει να δούμε ε, πολύ προσεκτικά τις συνδέσεις και γιατί δεν θέλουμε τα περιφερειακά μας ε, ε, αερολιμένε ή μικρέ εταιρείε να ζημιωθούν Τώρα, όσον αφορά κάποια άλλα θέματα για τη λάθος ορθογραφία κάποιων ονομάτων, συμφωνώ, αλλά για re rerouting και άλλους τρόπους μεταφορών. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με το rerouting ή με τη χρήση άλλων ε, τρόπων μεταφορών, μεταφορικών μέσων, αλλά να σας, να το, σας το αντιστρέψω. Και αν ήμουν στο Eurostar, ας πούμε, ένα πολύ γρήγορο τρένο, τι θα κάνατε, θα με βάζετε σε reroute στην Air France ή στην British Airways. Ρωτώ, γιατί θεωρούμε πως κάτι τέτοιο είναι εύκολο. Αυτομάτως μπορούν να ξαναμπούν σε ένα άλλο ε, χ αεροπλάνο αφόσον είναι διαθέσιμο. Όμως πρέπει κάπως περισσότερο να το σκεφτούμε, γιατί είναι κάπως αυθαίρετη αυτή η κατάσταση. Να δούμε ποιος πληρώνει τι και πώς θα γίνει ακριβώς. Γιατί σίγουρα από το Eurostar δεν με βάλανε σε κάποια πτήση. Κάποιες ε, μικρότερες παρατηρήσεις, γιατί εδώ υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες σε σχέση με την μη χρήση ε, των τομέων του, του ΑΛΕ. Κάποιος που, έχει κάνει μια σύμβαση με έναν πελάτη έχει όλες τις πληροφορίες. Η εταιρεία έχει κάνει οικονομικά μια καλή συμφωνία γιατί αυτό που θα πέσει ε, τελικά είναι οι φτηνές πτήσεις που επιτρέπουν ε, στους επιβάτες να υποφεληθούν. Αυτή θα είναι η συνέπεια. Πρέπει λοιπόν πολύ πολύ προσεκτικά να το σκεφτείτε αυτό. Και έπειτα, χειραποσκευή δεν είναι δική μας απόφαση, είναι εμπορική απόφαση. Και όσο αφορά τα duty free, τι είναι μια τσάντα duty free. Μπορώ να πάω να πάρω μια ζαβαλίτσα, να πάρω ένα ταγέρ και να μπορώ να το πάρω στο αεροσκάφος. Μα δεν είναι δική μας δουλειά να αποφασίσουμε ποια χειραποσκευή θα πάρει κανείς. Είναι οι αεροπορικές εταιρείε σε συνδυασμό με τα θέματα ασφάλειας και τι μπορεί να μπει και να κλείσει μέσα σε εκείνα τα ντουλαπάκια. Με την προϋπόθεση ότι οι επιβάτες θα ξέρουν τις πληροφορίες αυτές πριν να πληρώσουν το ειστήριό τους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό νομίζω. Αν γίνει λοιπόν, βέβαια υπάρχουν και ένα σωρό άλλες ψηλολεπτομέρειες, αλλά στη συνεδρία των σκιωδών θα συζητηθούν και θα δούμε πού θα καταλήξουμε. Όπως σας είπα, έχουμε κάποιες σοβαρές δυσκολίες με κάποια από τα ζητήματα. Αλλά ίσως να τα καταφέρουμε και να τα ξεπεράσουμε. Ίσως και όχι. Πάντως κάποια βασικά θέματα πρέπει να τα σκεφτούμε. Να ευχαριστήσουμε και πάλι τον εισηγητή για τη συμβολή του μέχρι στιγμής. Ευχαριστώ πολύ. Μιλήσανε όλοι οι σκιώδεις. Τώρα τα μέλη να ζητήσω ε, να μιλήσουν το πολύ τρία-τέσσερα λεπτά λεπτά γιατί έχουμε πολλούς υποψήφιους στον κατάλογο. Darlin, Mr. Cock, Mrs. Mr. Bradbourne. Anybody else wants to speak? Εκτός από τα ονόματα που αναφέρθηκαν υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει το λόγο. Α, και εγώ στο τέλος και κλείνει ο κατάλογος, εντάξει. Ωραία. Κύριος Γκρός. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και εγώ φυσικά θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή και τους συναδέλφους του για το έργο του, τους. Για μας το ΕΛΚ ο σημαντικός στόχος μας είναι να μάθουμε από τα διδάγματα του παρελθόντος ώστε η νομοθεσία να οδηγεί σε αποτελεσματική προστασία των ε, επιβατών. Αυτό θα πρέπει να είναι η απόλυτη προτεραιότητα όχι μονάχα να βελτιώσουμε τα δικαιώματα των επιβατών, αλλά να εξασφαλίσουμε και μία ασφάλεια δικαίου για τους επιβάτες. Επανέρχομαι σε αυτά που είπε η κυρία Φώστερ για τις αποσκευές. Αν μιλήσουμε μονάχα για ε, αποσκευές, για μια τσάντα γυναικεία ή μια τσάντα από ψώνια και είναι διαφορετική η βαλίτσα όπως το βλέπει ο ένας και όπως το βλέπει ο άλλος, αυτός, αυτό θα οδηγήσει σε ασάφεια και σε έλλειψη ασφάλειας για τους επιβάτες. Ενώ αν ξέρουμε ακριβώς ποια είναι, ποιοι είναι οι ορισμοί, θα βοηθήσει την ασφάλεια για τους επιβάτες. Για τις ανταποκρίσεις και γενικά την αντιμετώπιση υπάρχουν πολλές εταιρείες οι οποίες σέβονται τα δικαιώματα των ε, επιβατών τους δεν πρέπει να δώσουμε την εντύπωση ότι οι επιβάτες δεν ε, τους λαμβάνει κανείς υπόψη σε μια εταιρεία. Υπάρχουν εταιρείε με πολύ καλή εξυπηρέτηση των ε, επιβατών. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι σε, στις ε, αναπληρώσεις, στις ανταποκρίσεις, αυτός ο οποίος έρχεται καθυστερημένα να φέρει το βάρος, αλλά όταν η εταιρεία έχει καθυστερήσει το αεροπλάνο της, να μην φέρει το βάρος ο επιβάτης. Μεταξύ των τριών και των πέντε ωρών έχω ένα πρόβλημα. Όταν εμείς κάνουμε μια νομοθεσία και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταλήγει σε μια διαφορετική ρύθμιση. Εγώ πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να είναι αρμόδιο για τα θέματα αυτά. Δεν είναι το ε, δικαστήριο το οποίο πρέπει να νομοθετήσει τη θέση των κοινοβουλευτικών. Θα πρέπει να καθορίσει τις νομικές αρχές. Εγώ δεν πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να περιοριζόμαστε από τις αποφάσεις αυτές. Το δικαίωμα τώρα <clears throat> αγωγής. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να υπάρχει μια σαφής άρνηση των δικαιωμάτων και αυτό να οδηγεί σε δικαστικές διαδικασίες. Και πρέπει να υπάρχουν και λογικές αποζημίσει. Κάποιος ο οποίος παίρνει μια φθηνή πτήση δεν μπορεί να περιμένει μια πάρα πολύ ακριβή αποζημίωση. Θα πρέπει να υπάρχει και εδώ μια έννοια αναλογικότητα ώστε να μπορούν και οι επιχειρήσεις να λειτουργήσουν. Γι' αυτό λέμε για μένα το τι ακριβώς αποτελεί άρνηση των δικαιωμάτων των επιβατών είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να γίνει σαφέ ώστε να είναι και προ όφελο του επιβάτη η σαφήνεια που θα προκύψει. Τρία λεπτά κύριο Αλκαντράουι. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον συνάδελφο για τη δουλειά την οποία έκανε, τον κύριο Μπάχα. Όπως είπα εξ ονόματος της ομάδας μου υπάρχουν πάρα πολλά σημεία για τα οποία είμαι σίγουρος ότι θα πετύχουμε μια συμφωνία και θα είναι και ε, θετική η συνεργασία μας. Διότι πρόκειται για μια πάρα πολύ, ένα πολύ σημαντικό κείμενο. Ε, όλοι έχουμε ζήσει πολλές καταστάσεις, ε, αντιμετωπίσαμε προβλήματα τα οποία εμείς σαν πολιτικοί, πολιτικοί θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και να επιλύσουμε. Λοιπόν, ε, δεν θα κάνω, δεν θα πω πολλά πράγματα, θα περιοριστώ σε λίγα. Συμφωνώ με τον εισηγητή όταν λέει ότι θέλει να συζητήσει τα κατόφλια. Η Κομισιό ίσως να ήταν ιδιαίτερα περιοριστική. Αυτό, αυτή η καθυστέρηση πέντε ωρών ε, ίσως είναι μεγάλη και ο περιορισμός των αποζημιώσεων στην τιμή του εισιτηρίου ε, που είπε και η συνάδελφος από την είναι κάτι το οποίο μπορούμε να συζητήσουμε αλλά η τιμή του εισιτηρίου μπορεί να είναι μόνο ένα σημείο, ε, ένα κομμάτι της ε, ζημιάς που θα υποστείς λόγω της καθυστέρησης ίσως ε, μια σημαντική δουλειά που θα είχες ε, να μην ε, στεφθεί με επιτυχία και τέλος πάντων υπάρχει και ένα κόστος το οποίο δεν μπορεί να εκφραστεί αριθμητικά πάντα. Επίσης, η... θα... το, κατά πόσο, το, πώς θα εξετάσουμε το θέμα του χρόνου και του κόστους θα το ξαναδούμε όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει μια κάποια, ένας κάποιος παράγοντας ε, αβεβαιότητας. Διότι τι σημαίνει ε, απρόβλεπτες συνθήκες. Είναι πολύ ευρύ το πεδίο. Τεχνικά, ε, τεχνικές λεπτομέρειες, παραδείγματος χάρη, όπως μπορεί να χαρακτηριστούν απρόβλεπτες ε, συνθήκες. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ε, εξετάσουμε. Επίσης, ένα άλλο σημείο έχει να κάνει με την ενημέρωση και την διαφάνεια και ενημέρωση των ε, επιβατών. Τι προβλήματα μπορεί να υπάρξουν και τι βοήθεια μπορεί να ζητήσει ο επιβάτης. Τελευταία παρατήρηση αφορά τα εθνικά, τις εθνικές οργανώσεις, εθνικούς οργανισμούς για την ε, υποβολή παραπώνων τέλος πάντων. Ε, εδώ υπάρχουν προβλήματα, διότι δεν ερμηνεύουν όλοι οι οργανισμοί με τον ίδιο τρόπο την κατάσταση. Χρειαζόμαστε πιο αυστηρούς κανόνες και ίσως η Κομισιό ή και άλλοι ευρωπαϊκοί οργανισμοί θα πρέπει να εξασφαλίσουν ένα καλύτερο συντονισμό. Ο κύριος Βαντάμ για τρία λεπτά. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον εισηγητή σε όλες ε, αυτές τις συνθήκες ε, και τις περιστάσεις θα πρέπει σαν ε, ε, νομοθέτες, συνομοθέτες, να διευκρινίσουμε τα πράγματα. Θα πρέπει οι επιβάτες να ξέρουν ε, ποια είναι τα δικαιώματά τους και πιστεύω ότι ο κύριος Μπαχ συνεισφέρει σε αυτό. Ε, κάποια σημεία τώρα για τα οποία έχω κάποιες αμφιβολίες. Καταρχάς, ποιος είναι υπεύθυνο να βοηθήσει τους επιβάτες σε περίπτωση καταστροφής. Μόνο η αεροπορική εταιρεία μπορεί να το κάνει αυτό πώς θα ε, ρυθμιστεί σε συνεργασία με την ε, πολιτική αεροπορία, με τις τεχνικές υπηρεσίες. Αυτό είναι θέμα της αεροπορικής εταιρεία δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς τίποτα. Το πιο περίπλοκο θέμα είναι οι αποζημιώσεις και οι ε, καθυστερήσεις. Ε, ο εισηγητής μίλησε για, τις, για τρεις ώρες και πέντε ώρες. Τρεις εντάξει, αλλά πέντε ώρες ε, για πτήσεις, ε, για μεγάλες πτήσεις, ε, μεγάλες διάρκειας, εγώ θα έλεγα 6 με 7 ώρες, γιατί 5 ώρες για μεγάλες πτήσεις δεν είναι, δεν είναι, δεν είναι κάτι ασυνήθιστο. Συνήθως αυτές οι μεγάλες πτήσεις έχουν και μεγάλες καθυστερήσεις. Και θα έπρεπε να υπάρχει και ε, μια διαδικασία, ε, αν θέλετε, διαιτησίας ε, πολύ πιο απλή. Θα έπρεπε ο επιβάτης να έχει να αντιμετωπίσει μια διαδικασία απλή, να μην του περιπλέκουμε την κατάσταση. Τέλος πάντων, ε, και στο σημείο αυτό πιστεύω ότι, ότι ο εισηγητής τα έχει πάει καλά, υπάρχουν κάποιες εμβολίες, αλλά θα προχωρήσουμε. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Νομίζω ότι μπόρεσε ο, ο να καλύψει το μεγάλο χάσμα ανάμεσα στα δικαιώματα των επιβατών και των συμφερόντων των εταιριών. Ο στόχος μας δεν πρέπει να είναι να χρεοκοπήσουν οι εταιρείες αλλά να βελτιωθεί η ποιότητα των υπηρεσιών στους επιβάτες αεροπορικών εταιριών. Πρέπει επίσης να ληφθούν ιδιαίτερα υπόψη τα συμφέροντα των ατόμων με ειδικέ ανάγκες και γι' αυτό έχω καταθέσει αντίστοιχες τροπολογίες. Επίσης το να συνδέσουμε την αποζημίωση με την, την του εισιτηρίου αυτό είναι κάτι το οποίο αποφεύγει να κερδίσουν υπερβολικά λεφτά κάποια άτομα. Επίσης, στην περίπτωση της καθυστέρησης και οι επιβάτες είναι στη θέση τους, δεν μπορεί να αποφύγει την αποζημίωση η εταιρεία. Θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη. Ευχαριστώ. Κυρία Σενάλοβα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την ε, έκθεσή του. Είναι πολύ ε, σαφής η απόψη του, του. Ε, φαίνεται ότι έχει ξοδέψει πολύ χρόνο και τον ευχαριστώ που υιοθέτησε και προτεάσεις και από άλλες εκθέσεις όπου ασχολούμεθα με τα δικαιώματα των επιβατών. και ο εισηγητής και ο κύριος Αλκατράουι αναφέρθηκαν σε πολλά θέματα. Εγώ όμως θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για αυτές τις έκτακτες ή απρόβλεπτες συνθήκες. Και ευχαριστώ που μίλησε, που αναφέρεται ο κύριος Μπαχ στα θέματα αποζημιώσεων σε περίπτωση χρεοκοπίας της εταιρείας υπάρχουν, γίνονται διάφορες προτάσεις και για εναλλακτικέ ε, λύσεις. Ε, και στα θέματα της διαφάνειας ε, πρέπει να πω ότι υπάρχουν ε, πολλές ρυθμίσεις εδώ που μας βρίσκονται σύμφωνους, όμως αυτό το οποίο επίγει είναι ότι θα πρέπει να ενημερώνουμε σωστά και έγκαιρα τους επιβάτες. Αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει κάπου να αναφέρουμε περισσότερο και τα δικαιώματα των επιβατών. Και αυτά θα, τα δικαιώματα θα μπορούσαν να μπουν και στην κάρτα επιβίβασης κάπου. Αλλά τέλος αυτά είναι λεπτομέρειες. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Μπάχ για τη δουλειά που έκανα στην πρόταση αυτή. Πρέπει να σας πω ότι συμφωνώ με τα περισσότερα πόσα λέει. Κάποιες σύντομες παρατηρήσεις. Στην αρχή της συζήτησης αναφερθήκαμε στα θέματα των εθνικών αρχών, ε, των ρυθμιστικών αρχών αλλά πιστεύω ότι αυτό υπογραμμίζει το όλο θέμα, ανεξάρτητα τι θα γίνει με τον κανονισμό αυτό, γιατί μπορούμε να δώσουμε στους επιβάτες όσα ε, δικαιώματα θέλουμε, αλλά εάν δεν εφαρμοστούν σωστά, δεν έχει κανένα νόημα. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να ενδυναμώσουμε τον, τον ε, ρόλο των εθνικών ρυθμιστικών αρχών. Εγώ έχω διάφορα παράπονα από πλευρά ε, των, ψηφοφόρων μου για, τις, για τον τρόπο και για, τον, και για την, τις καθυστερήσεις όσον αφορά την επίλυση των διαφόρων προβλημάτων ε, ε, και φαίνεται ότι και ο Βρετανικός οργανισμός δεν είναι, δεν ε, είναι και αρκετά δυνατός αν θέλετε. Άρα εκεί πρέπει, κάτι πρέπει να κάνουμε. Επίσης αυτές οι έκτακτες ή οι ασυνήθιστες συνθήκες. Εδώ θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε λίγο το θέμα γιατί θα πρέπει να υπάρχει απόλυτη σαφήνεια για το τι αποτελεί έκτακτη περίσταση. Αλλιώς θα είναι και, και, λόγια όλα αυτά τα οποία λέμε. Η προσωπική μου εμπειρία είναι ε, στις που έχω ε, που παίρνω από τις Βρυξέλλες στην πόλη μου, τους τελευταίους μήνες έχω παρατηρήσει ότι έχει αυξηθεί ο ρυθμός των καθιστών ε, ακυρώσεων των πτήσεων για τεχνικούς λόγους, για βλάβια αεροσκάφους και θα πρέπει κάτι να κάνουμε αν αυτό συμβαίνει τακτικά. Κάτι πρέπει να γίνει και οι επιβάτες να μπορούν να παίρνουν μια κάποια σχετική αποζημίωση. Τρίτη παρατήρηση, Πρόεδρε. Και επανέρχομαι στην έκθεση του κύριου Τέιλορ. Ήθελα να πω ότι ίσως να ξέρουν και οι συνάδελφοι έχουν υποβληθεί τροπολογίες για για τις διευκολύνσεις ε, ε, για τα άτομα με σοβαρές αναπηρίες και θα ήθελα και ο κύριος Μπάχα να συμφωνήσει να υποβληθούν παρόμοιες τροπολογίες και στην δική του έκθεση αργότερα. Και η τελευταία παρατήρησή μου, τέταρτη και τελευταία, αφορά το θέμα των μεταφορών στα, αεροπλα... αεροδρόμια. Δεν, έχουμε... δεν ξέρω αν μπορούμε εμείς να αποφασίσουμε γι' αυτό, αλλά τέλος πάντων να νομοθετήσουμε. Αλλά ας πούμε εάν ε, χάσεις ε, την πτήση σου λόγω καθυστέρησης από άλλο αεροπλάνο και γιατί δεν γίνεται σωστά το transfer, ε, δηλαδή από τη μία πτήση στην άλλη, μέσα στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο, θα πρέπει κάτι να γίνει, γιατί πολλές φορές πολλές φορές ο επιβάτης χάνει την, την, την πτήση του γιατί ε, ο χρόνος που έχεις για να πάρεις την ανταπόκριση είναι πάρα πολύ ε, λίγος και όταν μιλάμε για αεροπλάνα, ε, ας πούμε, για αεροδρόμια μεγάλα όπως είναι το Παρίσι ή το Λονδίνο που περνάς από τη ζώνη Schengen σε ζώνη μη Schengen που πρέπει να περάσεις και έλεγχο διαβατηρίων κτλ εμείς μπορούμε να νομοθετήσουμε, αλλά από την άλλη πλευρά αυτός ο χρόνος ανάμεσα στις ανταποκρίσεις είναι μη ρεαλιστικός ε, και δεν γίνεται ό,τι και να πούμε εμείς. Τέλος πάντων, ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και κύριος κύριος Μπάχ να δεχτεί τις τοπολογίες. Πάρα πολύ σύντομα κύριε Κράμερ. Τόνισα τη σημασία του να υπάρχουν ανεξάρτητοι διαιτητές στην περίπτωση των σιδηροδρόμων έχουμε μια πολύ καλή εμπειρία και 90% μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν καθυστερήσεις ή όχι πραγματικές. Αυτό μπορούν να το κάνουν και οι αεροπορικές εταιρείες. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει ανεξάρτητη αρχή διαιτησίας στις επιχειρήσεις για να μπορούμε να αποφεύγουμε να φέρουμε όλα αυτά τα πράγματα στα δικαστήρια δεν επιλύονται ούτω ή άλλω. Εντάξει, από τη δική μου πλευρά λέει ο Μπράιν. Εγώ. Καταρχήν να πω ότι όποια συμπάθεια και να προ τι αεροπορικές εταιρείες εξαντλήθηκε στα αναρρύθμιτα ε, κτίρια των αεροδρομίων που έχουν περπατήσει κατά τη διάρκεια των ετών και επίσης είναι και ο τρόπος που σε αντιμετωπίζουν οι εταιρείε ε, δάυζου μου. Σου λένε, πά και τους ρωτάς μα γιατί ακυρώθηκε αυτή η πτήση και απλώς ε, ανασηκώνουν τους ώμους, δεν ξέρει ποτέ κάνει τίποτα. Και μετά τους λες μπορώ να μπορέσω λίγο να φρεσκαριστώ ή να μου δώσετε κάνα ψυχτικάκι και εκεί ε, σου λένε πω εδώ τώρα πρέπει να το εγκρίνει αυτό ο διευθυντής. Ε, πιστεύω ότι στην κατάρτισή τους θα έπρεπε να είναι υποχρεωτικό να γνωρίζουν απ' έξω και ανακατοτά τον κανονισμό 261 ή όποιο θα είναι το, το νούμερό του, εν πάση περιπτώσει, και έπειτα να δίνουν πληροφορίες στους, επιβάτε. επιβάτες. Δεν θα πρέπει να είναι απλά μια πινακίδα πίσω από ε, ένα μηχάνημα που πουλάει κοκακόλα που κανείς δεν μπορεί να το δει. Πρέπει να είναι στο check-in η σχετική επιγραφή Νομίζω πως το είδα μια φορά στην Νάπολη. Μπράβο στους Ναπολιτάνους λοιπόν. Και επίσης τι ενημέρωση δίνεται για τα δικαιώματα των, των, των επιβατών στα ηλεκτρονικά ειστήρια. Τίποτα. Μηδέν. Μηδέν. Τίποτα απολύτως. Λέει είναι ένα σωρό για το τι φόρο πληρώνεις, ένα σωρό νούμερα αναφορές με κεφαλαία γράμματα. Αλλά δικαιώματα των επιβατών. Τίποτα απολύτως πάνω στα ηλεκτρονικά ειστήρια. Και αυτό θα πρέπει να διορθωθεί. Και για τους κανόνες περί αποσκευών. Εγώ θέλω να πω μόνο πως δεν θα πρέπει να υπάρχουν εκεί διακρίσεις. Δεν μπορείς να έχεις ένα αεροδρόμιο που μπορεί να παίρνεις ε, μια συγκεκριμένη τσάντα ή στο άλλο όχι ή επειδή μια εταιρεία θέλει να πουλάει τα δικά της ε, duty free πάνω στο αεροπλάνο να μην επιτρέπει τις αγορές στο αεροδρόμιο κτλ. κτλ. Θα πρέπει να είναι όλα ομοιόμορφα, ιδιαίτερα όσον αφορά τις αγορές στους αερολιμάνες. Τώρα, τιμές των εισιτηρίων. Κάποιοι λένε ότι η αποζημίωση θα πρέπει να συνδέεται με τη τιμή του εισιτηρίου. Αλλά τι θα πει η τιμή εισιτηρίου? Τιμή του εισιτηρίου συν φορεί. Τιμή εισιτηρίου συν τα διάφορα επιπλέον κόστη τα ADP, αν δεν είσαι πολύ τυχερός ε, και προέρχεσαι από μια χώρα όπου υπάρχουν τέλη επιβατών ή 2-3 ευρώ που διαφημίζονται και που ποτέ κανείς δεν καταβάλει. Και έπειτα, η τιμή του εισιτηρίου σε καμία περίπτωση δεν αντικατοπτρίζει την δυσκολία που εσύ και ο κ. Αρκαντράη το ανέφερε, που εσύ οι επιβάτες έχουν περάσει. Την ταλαιπωρία αυτή δεν την επιληρώνουν. Θα πρέπει λοιπόν η υποζημίωση να συνδέεται με την ταλαιπωρία και όχι απαραίτητο με την τιμή του εισιτηρίου. Ελπίζω να μην πέσετε εσείς σε αυτή την παγίδα την οποία έχουν απλώσει κάποιες αεροπορικές εταιρείε ή μάλιστα οι εταιρείε αυτές για τις οποίες έχουμε τις περισσότερες καταγγελίες για το ότι η αποζημίωση θα πρέπει να συνδέεται με τη τιμή του ειστηρίου. Λοιπόν, το NB, e κατά τη γνώμη μου έχει αποτύχει με τον 201. Είναι ένα τσουβάλι ασυνέπειας. Και κάθε φορά κάνουν ε, λάθος, δεν θέλουν να υπάρχει σαφήνεια, δεν θέλουν να την προωθήσουν και κατά τη γνώμη μου δεν αντιπροσωπεύουν τους καταναλωτές όπως θα έπρεπε ε, και ενώ υποτίθεται ότι τους φροντίζουν και τους προστατεύουν. Θέλουμε λοιπόν να υπάρχει συνέπεια από τα NDB, να υπάρχει δηλαδή μια εναρμονισμένη προσέγγιση όσον αφορά την επιδίωξη αυτών των στόχων. Τέλος. Φόρος μαζέρ. Ανωτέρα βία. Εδώ πρέπει πολύ να σφίξουν τα πράγματα. Και μάλιστα ριζικά. Γιατί είναι παραθυράκι το οποίο χρησιμοποιούν αεροπορικές εταιρείε ώστε να αποφεύγουν τις υποχρεώσεις τους. Ας τα πούμε ξεκάθαρα. Και ο συμπεφωνημένος κατάλογος, κατάλογος που ανεφέρθη είναι ένας γιγάντιος γιγάντιο παραθύρι, παραθυράρα δηλαδή, για τις αεροπορικές εταιρείε ώστε να μην πληρώνουν αυτά που πρέπει. Και εγώ λοιπόν θα καταθέσω τροπολογίες που θα περιορίζει την ανωτέρα βία σε δύο-τρία σημεία. Και εκτιμώ τις προσπάθειες του, του εισηγητή για την ε, ανωτέρα βία και νομίζω πως ο Τζόρτζ δεν, δεν έχει πάει αρκετά μακριά. Οτιδήποτε είναι τεχνική φύσης δεν είναι ανωτεραβία, είτε είναι ε, εξάρτημα, παραεξάρτημα, πρώτο, ε, καινούριο, μεταχειρισμένο κτλ. Ο επιβάτης αυτό που ξέρει είναι ότι δεν του δίνεται αποζημίωση διότι η υδραυλική βαλβίδα της δεξιάς, ε, του, του δεξιού κινητήρα ήταν ένα ελάττωμα από τη μάνα του αεροπλάνου ή όχι. Τι τον ενδιαφέρει τον επιβάτη αυτό. Αυτό τον ε, ενδιαφέρει αν θα πάει στη δουλειά του ή όχι. Ανώτατη, ανωτέρα βία είναι τα ηφαίστεια, η κακοκαιρία. Ε, από εκεί και πέρα πραγματικά είναι υπερβολικό. Και αυτή τη γραμμή θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Τούτον τον Τζόρτζ έχει φτιάξει εξαιρετική έκθεση είναι μια πολύ καλή βάση για να συζητήσουμε και νομίζω πως η θέση σου και η κατεύθυνσή σου είναι απόλυτα σωστή. Γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής θα πρέπει να θυμόμαστε τι θέλουμε να κάνουμε με αυτήν εδώ την οδηγία. Δικαιώματα επιβατών, όχι δικαιώματα αεροπορικών εταιριών, ε, δικαιώματα επιβατών. Ο κύριος Φόλζεν από την Κομισιόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την έκθεσή του που καταδεικνύει την καλή γνώση όλων αυτών των θεμάτων και για τις καλές σχέσεις που είχε με την Κομισιόν. Το σχέδιο έκθεσης αναγνωρίζει δύο από τις προτεραιότητες που διείπαν το έργο της Κομισιόν. Μεγαλύτερη νομική ασφάλεια και καλύτερη εφαρμογή. Χαιρετίζουμε επίσης το γεγονός ότι το σχέδιο έκθεσης διευκρινίζει και αναπτύσσει περισσότερο ορισμένα θέματα όπως είναι οι αλλαγές τρομολογίου ε, μεταξύ των οποίων και η πτήση που φεύγει πιο νωρί ή όταν χάνει επιβάτης την πτήση επειδή φεύγει πολύ νωρί. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον εισηγητή για το γεγονός ότι εντοπίζει προβλήματα σε σχέση με την εφαρμογή του κανονισμού σε ανταποκρίσεις που τις χάνει κανείς λόγω καθυστέρησης. Το σχέδιο έκθεσης πιστεύουμε κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά νομίζουμε ότι είναι απαραίτητο να αξιολογηθούν όλες οι πτυχές της προτινόμενης λύσης. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε επίσης τον εισηγητή γιατί ανέπτυξε περισσότερο την ιδέα της πολυτροπικής μεταφοράς όταν συνδυάζεται η αεροπορική πτήση με μια μεταφορά συντροδομική. <clears throat> Είμαστε ανοιχτοί επίσης και με την ιδέα του να μειώσουμε την καθυστέρηση στην πίστα σε λιγότερο από πέντε ώρες. Αλλά συγχρόνως πιστεύουμε ότι οι τροπολογίες εκφεύγουν από τον στόχο του να εξασφαλίσουμε μια σωστή ισορροπία μεταξύ των συμφερόντων των επιβατών και του οικονομικού αντικτύπου στον αεροπορικό τομέα που είναι και ένα από τα θέματα που ενδιαφέρουν την Κομισιόν. Πιστεύουμε λοιπόν ότι ορισμένε από τις τροπολογίε έχουν αντιπαραγωγικό αποτέλεσμα για τους ίδιους επιβάτες. Παραδείγματο χάρη. Θα αναφέρω τα εξή θέματα. Πρώτα απ' όλα το κατόφλι των τριών ωρών καθυστέρηση για να πάρει ο επιβάτης αποζημίωση. Πιστεύουμε ότι τρει θα οδηγήσουν το όριο των τριών ώρων, θα οδηγήσει σε περισσότερε ακυρώσει πτήσεων. Μια καθυστέρηση για μια πτήση έχει αντίκτυπο στις επόμενε πτήσει με το ίδιο αεροσκάφο. Οι αεροπορικέ εταιρείε πρέπει να δώσουν επομένω αποζημίωση όχι μόνο στον επιβάτη τη καθυστερημένης πτήση, αλλά και στου επιβάτε των μεταγενέστερων πτήσεων με το ίδιο αεροσκάφο, διότι και αυτοί θα καθυστερήσουν. Η αποζημίωση λοιπόν είναι τέτοια που οδηγεί στην ακύρωση μια ή δύο πτήσεων για να μπορέσει η εταιρεία να ξαναλειτουργήσει σωστά το χρονοδιάγραμμά της και οι επόμενες, εταιρεί... πτήσεις να είναι έγκαιρες. Αλλά για τους επιβάτες η ακύρωση είναι χειρότερη από την καθυστέρηση γιατί η δυνατότητα εναλλακτική πτήσης και διαδρομής δεν είναι πάντα εξασφαλισμένη. Γι' αυτό η Κομισιόν προτείνει μεγαλύτερα χρονικά κατόφλια. Το δεύτερο σημείο όπου ο εισηγητής προτείνει να αυξηθεί με έμεσο τρόπο το ποσό της αποζημίωσης. Προτείνει ο εισηγητής η αποζημίωση να περάσει από τα 200 ευρώ σε 300 ευρώ <clears throat> για πτήσεις κάτω από τα 1500 χιλιόμετρα. Και από 400 ευρώ σε, να μειωθεί σε 300 ευρώ για πτήσεις μεταξύ 1500 χιλιόμετρα και 3500 χιλιόμετρα. Αλλά 72% των επιβατών πετάνε σε πτήσεις κάτω από 1500 χιλιόμετρα. Αυτό το 20 και επίσης 21% των επιβατών πετάνε μεταξύ 1500 χιλιόμετρων και 3.500 χιλιόμετρων. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι ότι κατά μέσο όρο οι αποζημιώσεις αυξάνονται. Σε ό,τι αφορά τις προτινόμενες τροπολογίες <clears throat> για τις έκτακτες περιστάσεις. Νομίζουμε ότι η τροπολογία αυτή ξεπερνάει, μάλλον αποκλίνει από την ε, απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, αποκλείοντας περιπτώσεις στις οποίες δεν έχουν καμία, κανένα έλεγχο οι αεροπορικές εταιρείες. Τέλος, σε ό,τι αφορά την πτώχευση των αεροπορικών επιχειρήσεων. Κατανοεί η Κομισιόν τις ανησυχίες του εισηγητή, αλλά πιστεύει ότι μια υποχρέωση για τις εταιρείε να δίδουν εγγυήσει επαναπατρισμού μέσω ενός ε, ταμείου, αυτό πάει πολύ μακριά. Γιατί με τον τρόπο αυτό διπλασιάζεται το κόστος για τις επιχειρήσεις αυτού του κανονισμού. Είναι και δυσανάλογο προς την κλίμακα του προβλήματος τα τελευταία 10 χρόνια 0,07% όλων των ταξιδιών επηρεάστηκαν από τέτοιες φτωχεύσεις και μόνο 12% των επιβατών που εμπλεκόταν βρέθηκαν χωρίς δυνατότητα επιστροφής. Η Κομισιόν πιστεύει η Κομισιόν πιστεύει ότι αυτό το θέμα πρέπει να ρυθμιστεί επί τη βάση ανακοίνωσή τη του Μαρτίου αυτού του έτους η οποία έχει μεταφραστεί σε συγκεκριμένες δράσεις, όπως πιο σωστή παρακολούθηση της ε, χρηματοπιστωτικής υγείας των ε, αεροπορικών επιχειρήσεων και συζητήσεις με τους εμπλεκόμενους για να υπάρξει δημιουργία ενδιάμεσων προϊόντων. Η Κομισιόν πρότεινε επίσης να υπάρξει και ανάπτυξη σχεδίων Αντιμετώπιση έκτακτων συνθηκών στα αεροδρόμια που αντιμετωπίζουν περιπτώσεις όπου έχει υπάρξει πρόβλημα πτώχευσης μιας επιχείρησης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εντάξει λέει ο Μπράιν, πολύ καλά. Κύριε Ισηγητά, αν θέλετε να απαντήσετε σε όλα αυτά. Ευχαριστώ, λέει ο κύριος Μπαχ. Πάρα πολλά θα έπρεπε να πω αλλά σε λίγα λεπτά θα σταθώ μοναχά σε ορισμένα σημεία. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για την υποστήριξη που μου έχουν δώσει. Είναι καθυσυχαστικό όταν του λένε συναδελφοί του σε κανένα ότι κινείται σε σωστή κατεύθυνση και θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για την εμπιστοσύνη που μου δίνουν. Βέβαια υπάρχουν και κρίση, επικριτικές στάσεις. Ακόμα και αυτές οι επικρίσεις τις λαμβάνω πολύ στα σοβαρά και σίγουρα θα τις λάβω υπόψη στην εκπόνηση της έκθεσης, στην τελική μορφή. Ξεκινήσω με το θέμα της πτώχευσης των αεροπορικών εταιριών. Υπάρχει καταρχήν ένα πρόβλημα σε σχέση με την ισορροπία. Με αυτούς οι οποίοι πετάνε με, κάποιους, με κάποια ταξίδια που, συμπεριλαμβάνουν, που είναι συνολικά συμπεριλαμβάνουν ταξίδι και ε, στέγαση και αυτούς που πετάνε μεμονωμένοι. Εδώ είναι πολύ δύσκολο να εξασφαλίσουμε τη σωστή ισορροπία γιατί δεν έχουμε μοναχά τους ε, επιβάτες οι οποίοι ε, τους αφήνει η αεροπορική εταιρεία στη, σε κάποιο άσχετο σημείο αλλά και αυτούς που δεν έχουν φύγει καν από το σπίτι τους γιατί δεν έχουν προλάβει να πετάξουν. Η Κομισιόν ζητά να υπάρξει μια υπεύθυνη στάση από τα κράτη-μέλη για τα θέματα αυτά και όλοι ξέρουν ότι τα κράτη-μέλη ε, θεωρούν ότι οι επιχειρήσεις πολλές φορές δεν μπορούν να πληρώσουν και δεν τις πιέζουν. Αυτό δεν επαρκεί. Νομίζω ότι ο πρόεδρος μας τα είπε πολύ ωραία. Έχει εκφράσει πολύ έντονα και ενεργητικά τα θέματα αυτά. Οι επιχειρήσεις λένε πάντα για να πετύχουν το καλύτερο image ότι πρώτα απ' όλα είναι η ασφάλεια και μετά έχουν μια σωρία από τεχνικά προβλήματα. Εδώ υπάρχει μια εγγενής αντίφαση. Είτε θέλει κανείς να έχει το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας ή αλλιώς λέει ανά πάσα στιγμή μπορούμε να έχουμε τεχνικά προβλήματα. Δεν μπορεί να το λέει αυτό μια επιχείρηση και να χρησιμοποιεί τέτοια παρατηράκια. Ε, συνολικά πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να βρούμε κάποιε λύσει μαζί με του συναδέλφου. Θέλω να πω κάτι επίση για το θέμα τη αναλογικότητα, όπω ανέφερε ο πρόεδρο μα για τα θέματα των εισιτηρίων και των αποζημιώσεων. Είναι σαφές εδώ ότι δεν μιλάμε σε μια προσαρμογή σε σχέση με το ποσό που καταβλήθηκε από τον ε, καταναλωτή έχει αποφασιστεί και έχει εδρεωθεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ότι πρόκειται για μία αποζημίωση για την ε, ταλαιπωρία του επιβάτη και όχι για ένα ποσό που συνδέεται με το εισιτήριο γιατί ο επιβάτης θα πρέπει να στεγαστεί, να φάει επομένως και χάνει τον χρόνο που του είναι πολύτιμος επομένως εδώ δεν μπορεί κανείς να το συνδέσει αυτό με το εισιτήριο πρέπει να είναι ένα ποσό το οποίο είναι απόλυτο και κατά αποκοπή. Επομένως υποστηρίζω και τονίζω ότι η αποζημίωση πρέπει να είναι ενιαία. Για τα χρονικά όρια. Τρεις ώρες ή πέντε ώρες. Αυτά μπορούμε να τα συζητήσουμε. Ο Ματιού έφυγε. Αλλά θα του πω, θέλω να του πω ότι δεν μας έχει γονατίσει μέσα σε εισαγωγικά η απόφαση του δικαστηρίου. Εγώ δεν συμφωνώ με την Κομισιόν, θαυμάζω την στάση της ίσως, αλλά θέλω να τονίσω ότι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξέρουν ποια είναι τα δικαιώματά τους με την ομολογία του δικαστηρίου και θα είναι σημαντική υποχώρηση αν μειώσουμε τα υφιστάμενα δικαιώματα των επιβατών και περάσουμε από τις 3 στις 5 ώρες ως κατόφλι. Και για τις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, αυτά που ελέγχθηκαν είναι σωστά. Υπάρχουν πολλά αεροδρόμια όπου αντιμετωπίζονται σωστά τα θέματα αυτά και νομίζω ότι πρέπει και οι εταιρείε να παίζουν κάποιο ρόλο για να βελτιωθεί καλύτερα η εξυπηρέτηση στα αεροδρόμια. Και αυτό μας δώσει καλύτερα αποτελέσματα. Αυτά λοιπόν. Νομίζω ότι έχω καλύψει τα πιο σημαντικά θέματα και φυσικά τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε και με όλους τους συναδέλφους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μπάρκ. Θα ήθελα να σας θυμίσω, γιατί ξέρω πως δεν, υπάρχουν και ε, δεν θα υπάρχουν πολλές τροπολογίες. 3 ε, Οκτωβρίου είναι η προθεσμία υποβολής τροπολογιών στις 12. 3 Οκτωβρίου στις 12. Και αυτές τις ε, τροπολογίες θα τις εξετάσουμε στις 4 Νοεμβρίου και θα ψηφίσουμε στις 14 Νοεμβρίου στην Επιτροπή Μεταφορών. 3 Οκτωβρίου λοιπόν προθεσμία υποβολή τροπολογιών, 4 Νοεμβρίου, Νοεμβρίου εξέταση τροπολογιών και 14 Νοεμβρίου ψηφοφορία. Σας ευχαριστώ πολύ και τώρα περνάμε στο επόμενο θέμα. Εξακολουθούμε με την μάχη για την πολιτική αεροπορία. Εδώ έχουμε η συγγήτρια την κυρία Ντεβεράκ. Κριστίν, έχεις το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ψηφίσουμε αύριο για την έκθεση ε, αυτή που αφορά την αναφορά περιστατικών στην πολιτική αεροπορία. Ο διπρόεδρος διακόπτη, με συγχωρείτε λίγο, αλλά όποιοι φεύγουν να φεύγουν εισήχως ώστε να συνεχίσουμε εμείς τις εργασίες μας εδώ. Σα ευχαριστώ για τις πολυάριθμες τροπολογίε που έχουν κατατεθεί, 83 στον αριθμό και που οι περισσότερε επιτρέπουν να καταστεί το κείμενο πιο πλήρε και πιο σαφέ, έτσι ώστε ο καθένα να έχει ε, την ίδια ερμηνεία. Είναι σημαντικό να έχουμε ένα σαφέ κείμενο το οποίο να μπορεί εύκολα να εφαρμοστεί από τι διάφορε οργανώσει τα κραταμέλη και την Ίζα έτσι ώστε να έχουμε και επίτευξη των στόχων μας. Όπως το εξήγησα και στην προηγούμενη ανταλλαγή απόψεων και όπως το επιθυμούσε και η πλειοψηφία των συναδέλφων που πήρε το λόγο τότε, προσπάθησα να διατηρήσω τους στόχους του σχεδίου κανονισμού, καθιστώντας πιο ευέλικτη αυτό το κανονισμό, αλλά και πιο δεσμευτικό όσον αφορά την εμπιστευτικότητα και την προστασία των πληροφοριών που ανταλλάσσονται. Κοίταξα λοιπόν με προσοχή όλες τις τροπολογίες και υπέβαλα ε, στους σκιώδεις 7 συμβαστικές που όλες υποστηρίχθηκαν από τις διάφορες πολιτικές ομάδες. Το κείμενο που θα ψηφιστεί αύριο θεωρώ πως είναι ισορροπημένο και θα μπορούσε να αποτελέσει μια εξαιρετική βάση για διαπραγματεύσεις εν ώψη του τριλόγου τριμερούς διαλόγου. Ε, πρόκειται για ένα σύνολο μέτρων που στόχο έχει τη δημιουργία ενός πνεύματος μιας κοινή νοοτροπίας ε, ε, κουλτούρας. Δεν χρειάζεται να επεκταθώ περισσότερο για αυτό το θέμα σήμερα, αλλά είναι πολύ σημαντικό το προσωπικό της πολιτικής αεροπορίας να μπορεί να αναφέρει ένα περιστατικό χωρίς να φοβάται πώς θα έχει να αντιμετωπίσει αντίπεινα ιεραρχικά ή νομικά και αυτό μόνο και στόχο να ενισχυθεί η ασφάλεια. Πρόκειται και μια εναρμόνιση προς τα πάνω και γι' αυτό μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι. Οι συμβαστικέ, επί των οποίων θα ψηφίσουμε αύριο, επιτρέπουν περισσότερη ευελιξία στη διαδικασία και επιτρέπουν επίσης στις μικρές οργανώσεις, αναπερίπτωση και στη συμφωνία με τις αρμόδιες αρχές, να φτιάχνουν απλοποιημένα συστήματα για τη συλλογή, την επεξεργασία και την ανάλυση των δεδομένων. Το κείμενο θα επιτρέψει επίσης την αποσαφήνιση του ρόλου καθενός από συμμετέχουν στο σύστημα αναφορών περιστατικών, δηλαδή ε, προσωπικό, κρατημέλη, ε, ΕΑΖΑ, όλοι θα έχουν συγκεκριμένο ρόλο και υποχρεώσεις μέσα, μέσα μάλλον από αυτό το μηχανισμό και έτσι θα ενισχυθεί η ασφαλής ανταλλαγή στοιχείων ώστε να μπορούν να ληφθούν σύντομα και ε, ταχαίως διορθωτικά μέτρα εφόσον εντοπίζεται κίνδυνο για την ασφάλεια. Καλύτερη συλλογή στοιχείων, καλύτερη ανταλλαγή αυτών, καλύτερο εντοπισμό των κινδύνων ε, για, για την εναέρια ασφάλεια. Σε αυτά όλα αναφέρεται το κείμενο επί το οποίο θα ψηφίσετε αύριο το πρωί και μπορεί να ενισχύσει πραγματικά ένα ε, δραστήριο και σύστημα εντοπισμού κινδύνου ε, για τις αεροπορικές μεταφορές και να βελτιωθεί ο μηχανισμός πρόληψης ενώ αυξάνεται η κυκλοφορία των... στην πολιτική αεροπορία. Ευχαριστώ τους σκιώδες που συνεργάστηκαν για να βρούμε μια ισορροπία και πρόεδρε αν και είμαι συγχύτρια νομίζω πως ε, κατάφερα να μείνω στα τρία λεπτά. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Λάικφρυ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και την εισηγήτρια. Ήταν πολύ ευχάριστη συνεργασία. Πάντοτε είναι καλή βέβαια συνεργασία. Αλλά τέλος πάντων. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Πάντοτε είναι καλό το κλίμα ανάμεσα στην κυρία Ντεβεϊράκα και σε μένα. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι λίγο πολύ έχουμε την ίδια θέση δεν υπάρχει κάτι να γελάτε. Μία αρχή που ήταν πάρα πολύ σημαντική και για τους δυο μας είναι ότι θα έπρεπε να συμμετέχουν και οργανισμοί που είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η ΆΣΑ, παραδείγματος χάρη, αυτό ήταν πάρα πολύ καλό. Ε, θα πρέπει η ΆΣΑ να μπορεί να εκτελεί τα καθήκοντά της. Και η δεύτερη ερώτηση που ήταν ένα πολύ σημαντικό θέμα για όλους μας είναι ότι θα έπρεπε να έχουμε ένα γενικό σύστημα για οτιδήποτε πετάει. Αυτό υπήρχε και τώρα νομίζω ότι υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στα περίπλοκα αεροπλάνα και στα πιο απλά. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Και υπάρχουν και βέβαια και άλλα θέματα τα οποία δεν καλύπτονται από τις 7 συμβαστικές ε, τροπολογίες. Η σοσιαλιστική ομάδα θα υποστηρίξει τις ε, συμβιβαστικές τροπολογίες αλλά και, οι άλλ, και τις άλλες ε, τροπολογίες της κυρίας Ντεβεϊράκ, τόσο από μία. Και η κυρία Ντεβεϊράκ ε, δέχεται τις δικές μας τροπολογίες, άρα πρόκειται για μια έκθεση πολύ ισορροπημένη. Γιατί ο στόχος, μας, ο στόχος όλων μας είναι να εξασφαλίσουμε ένα υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας στις ε, αεροπορικές μεταφορές. Ευχαριστώ κυρία Ντεβεϊράκ και ευχαριστώ και τους άλλους συναδέλφους. Ήτανε εξαιρετική η συνεργασία μεταξύ όλων μας και ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου επιτρέψατε να μακρηγορήσω σήμερα. Ναι, ναι, ε, ε, το ήξερα ότι μιλούσατε τόσο καλά αγγλικά, γι' αυτό σας άφησα, για τους φιλελεύθερους. Αγαπητοί συν κύριος κατσίνα ε, ε, κύριε Πρόεδρε, κυρία Εισηγήτρια, πραγματικά ήταν ευχαρίστηση η συνεργασία με την κυρία Ντεβεϊράκα. Έχουμε ένα τεχνικό κείμενο που αφορά ε, διάφορες δραστηριότητες και εκφράζει διάφορα, διάφορες ομάδες συμφερόντων. Πολλά ακούστηκαν για το πώς θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε τον κανονισμό. Ακούστηκαν απόψεις για, την, για το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού, για την συμπερίληψη συμπερίληψη τη ΙΑΣΑ, για τη συμπερίληψη των αποκλεισμό κάποιων τομέων τη πολιτική αεροπορία. Όμω παρόλα αυτά υπήρχε ε, γενικότερη συμφωνία για τη συμπερίληψη πολλών ε, σημείων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον κανονισμό. Η η συγγήτρια αποτέλεσε ε, την ε, καθοδηγητική δύναμη, αν θέλετε, ακόμα και στις ε, συμβαστικές τροπολογίες τις οποίες η ομάδα μου υποστηρίζει. Η βασική μας ανησυχία ήταν ότι οι μικρότερες αεροπορικές εταιρείες στην, στις αεροπορικές μεταφορές θα αντιμετώπιζαν ένα δυσανάλογο φορτίο υποχρεώσεων δεν είμαστε τελείως ε, δυσαρεστημένοι με το τελικό κείμενο, αλλά πιστεύω ότι το τελικό κείμενο που θα εξετάσουμε αύριο θα αποτελέσει μια πάρα πολύ καλή βάση για τον τρίλογο. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για την συνεργασία που είχαμε μέχρι τώρα. Ευχαριστώ κυρία εισηγήτρια, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ ο κύριος, η κυρία Λίχτεμπεργκερ για τους πράσινους. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, την εισηγητρία, συγγνώμη. Είχαμε μια πλήρη συζήτηση μεταξύ μας και νομίζω ότι οι προτάσεις της είναι πολύ θετικές. Έχουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό καταφέρει να καταλήξουμε σε συμφωνία για ορισμένε τροπολογίες οι οποίες <clears throat> θα μπορέσουν να παρουσιαστούν στην τελική τους διατύπωση ω συμβαστικέ τροπολογίε. Πρόκειται για ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα και νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε σε ένα πολύ σημαντικό βήμα ώστε να έχουμε τη δυνατότητα μεγαλύτερη πρόληψη σε θέματα ασφάλεια, κάτι το οποίο έχει παραμεληθεί στο παρελθόν και γι' αυτό η ελπίδα μου είναι στην ψηφοφορία να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια σωστή πρόταση η οποία θα οδηγήσει σε ουσιώδεις βελτιώσει και έτσι ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μπορέσουμε να δώσουμε τη δική μας συμβολή για τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ κυρία, κυρία Φώστα. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και την συγγήτριά μας, την Κριστίν Ντεβεράκ για το έργο το οποίο έχει κάνει. Και εγώ συμφωνώ με αυτά που είπε η προλαλή η κυρία Λίχτεμπεργκερ. Έχουμε πετύχει μια μεγάλη συνένεση και μπορούμε να έχουμε μια πολύ καλή ψηφοφορία αύριο. Είναι κρίμα γιατί έχουν περάσει, πριν έχουν περάσει 10 χρόνια από τότε που εισήχθη η υποχρεωτική αναφορά των περιστατικών και υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη τα οποία συμμορφώνονται και υπάρχουν πολλά κράτη-μέλη τα οποία δεν έχουν <clears throat> συμμορφωθεί με τα θέματα αυτά. Εγώ δεν αναφέρομαι τώρα στην Κροατία που έχει μόλις γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά είναι πολλά τα κρατημέλη τα οποία δεν έχουν θεσπίσει τις απαραίτητες διαδικασίες για ένα σύστημα υποχρεωτικής αναφοράς των περιστατικών μιλάμε για την εφαρμογή και την αστυνόμευση. Είναι καλό να έχουμε οδηγίε, αλλά όταν δεν εφαρμόζονται, αυτό δεν μα οδηγεί πουθενά. Είναι λοιπόν σκόπιμο να το τονίσουμε και πάλι, όπω λέει η κυρία Ντεβεράκ, μια σωστή, ένα σωστό κλίμα, μια σωστή κουλτούρα για τα θέματα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά και είναι κρίμα το να μην μπορούμε σε πολλά κράτη-μέλη να έχουμε ένα εθελοντικό σύστημα παράλληλα με το υποχρεωτικό σύστημα. Κάτι το οποίο ισχύει στο Ηνωμένο εδώ και 20 χρόνια. Αυτό είναι ένα σύστημα που έχουν θεσπίσει οι αεροπορικές εταιρείες, επομένως δεν τηρεί τι προποθέσει για υποχρεωτικό. Αλλά τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εξετάσουν και αυτή τη δυνατότητα. Χρειάζεται λοιπόν να υπάρξει μεγαλύτερη σαφήνεια γιατί κάποια κράτη-μέλη δίδουν ε, πλήρεις ε, αναφορές ενώ κάποια άλλα δεν φτάνουν στο απαραίτητο σημείο. Θα ήταν χρήσιμο να καταλήξουμε σε μία συνένεση, μία συμφωνία μεταξύ των διαφορετικών νομικών συστημάτων στα διάφορα κράτη-μέλη. Γιατί τελικά είναι θέμα πολιτισμικό. Υπάρχουν κάποια κράτη όπου δεν θέλουν να ρίξουν το φταίξιμο σε κάποιον όταν αναφέρεται κάποιο περιστατικό. Ενώ σε άλλες χώρες θεωρείται αυτόματα ότι όταν λέτε για ένα περιστατικό κάποιος θεωρείται αυτόματα ότι είναι ένοχος και πρέπει να αποδείξει την αθότητά του. Δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο, θέλουμε να κάνουμε το αντίθετο απλώς να έχουμε την πληροφορία για το τι έχει γίνει. Αλλά θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για να υπάρξει ένα ομοιόμορφο σύστημα στα κράτη-μέλη και η ομάδα μας θα υποστηρίξει την κυρία Ντεβεράκ. Υπάρχει μόνο μια συμβαστική τροπολογία που θα υποστηρίξουμε, το ξέρει η κυρία Ντεβεράκ. Όλες τις άλλες τις υποστηρίζουμε, αλλά δεν θα δεχτούμε τη συμβαστική τροπολογία για αυτό, η οποία αφορά τον ορισμό της βαριάς αμέλειας. Όλες τις άλλες τις υποστηρίζουμε και θα ευχαριστήσω ιδιαίτερα την εισηγητρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, συγχαρητήρια κυρία Βεϊράκα. Η, η έκθεση σας, όπως θα περίμενα εξάλλου από σας, είναι εξαιρετική, είναι ακριβής και δεν με εκπλήσει το γεγονός ότι ε, έγινε αντικείμενο γενικύτερης ε, συνένεσης και ε, σίγουρα στη συνεργασία με τους άλλους συναδέλφους καταλήγουμε σε καλές απόψεις. Διαφωνώ μόνο σε ένα σημείο κύριε Πρόεδρε και εδώ συμφωνώ με την κυρία που μίλησε προηγουμένως. Δηλαδή εγώ στην τροπολογία υπαριθμών 90 αναφέρομαι στην, στις επι, σοβαρές Απόλυ, ε, αμέλειες, αμέλεια. Υπάρχουν δύο έννοιες που δεν μπορούμε να τις αναμίξουμε όσον αφορά την ευθύνη. Το ένα είναι ο δόλος και το, η ευθύνη. Όλα αυτά δεν μπορούν να ανακατευθούν και δεν είναι σωστή η πρόταση, κατά την άποψή μου, ε, η πρόταση της Κομισιόν, ούτε η τροπολογία 21 της κυρίας Ντεϊβιράκ και ούτε το υβρίδιο, το οποίο είναι το αντικείμενο της ε, συγχώνευσης των δύο. Και δημιουργούμε ένα νομικό ε, τέρας, τέλος πάντων, το οποίο ε, δεν μας οδηγεί πουθενά. Ο δόλος δεν μπορεί να εμφανιστεί σε βαθμίδες αν θέλετε. Ή υπάρχει δόλος ή δεν, δεν υπάρχει. Τώρα, από εκεί και πέρα θα μπορεί να γίνει, μπορούμε να λάβουμε υπόψη μας, ε, ας πούμε, την ε, παράληψη. Η παράληψη, ναι, και μιλήσουμε τώρα για νεοπολιόντιο κώδικα κτλ. κτλ. Το παρελθόν σε μια έκθεση που αφορούσε τα πλοία. Εκεί αναφερόμαστε ε, στην, στην σχέση δόλου και αμέλειας ή παράληψης γιατί το πρόβλημα ήταν να μην πληρώνουν τα πλοία για να μπορούν να μολύνουν. Εδώ όμως δεν μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Ξέρω ότι η κυρία Ντεβέιρακ στην έκθεσή της είχε τις καλύτερες προθέσεις και το έκανε γιατί δεν ήθελε να, να δώσει ευθύνες εκ των προτέρων και θα ήθελε να διατηρήσει διατηρήσει μια κάποια ε, ισορροπία. Όμως εδώ δεν μπορούμε να συνδέσουμε τον δόλο με την αμέλεια, είτε είναι μεγάλη ή μικρή αμέλεια. Δηλαδή θα πρέπει αυτά να τα ε, ξεκαθαρίσουμε. Σε αυτό το σημείο διαφωνώ κυρία, κύριε Πρόεδρε και κατά τα λοιπά η κυρία Ντεβεϊράκ με βρίσκει απόλυτα σύμφωνα σε αυτά τα οποία λέει. Ευχαριστώ. Ξέρω ότι εμείς στην Επιτροπή Δυναμική ε, περιμέναμε να μας στείλουν κάποια γνωμοδότηση. Μπορούσαν να το κάνουν, το επιθυμούσαν, αλλά δεν το έκαναν. Εγώ θέλω απλά να πω ότι ιδιαίτερα όσον αφορά τα ατυχήματα υπάρχει αυτό το πρόβλημα στην Ευρώπη ότι με τα διαφορετικά δυναμικά συστήματα. σε ορισμένες χώρες η αστυνομία αναλαμβάνει και μετατρέπεται σε ποινική έρευνα πριν να έχει καθοριστεί το αίτιο του ατυχήματος. Δεν έχω απάντηση για το πώς μπορεί κανείς να το παρακάμψει αυτό, αλλά γιατί είναι διαφορετικά τα συστήματα. Είναι όμως ένα πρόβλημα και πρέπει κάποια στιγμή να μπορέσει να λυθεί. Έχω τον κύριο Κορνέλης από την Κομισιόν. Σύντομα παρακαλώ. Ναι βεβαίως. Εδώ εμείς είδαμε και φάνηκε αυτό από τη συζήτηση ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν μπορεί ούτε η Κοινωνική Επιτροπή να το λύσει. Είναι ένα πρόβλημα που έχει να κάνει με την κατανομή της ευθύνη. Έχουμε διαφορετικές διατάξεις για την ε, ποινική δικαιοσύνη στα κράτη-μέλη και διαφορετικά δικαιώματα πρόσβασης και ε, μήνυσης για τα θέματα αυτά. Οπότε δεν είναι εύκολο αυτό να λυθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι, λέει ο Πρόεδρος, και αυτός είναι και ο λόγο γιατί είναι πολύ δύσκολο αυτό να επιληθεί σε μια γνωμοδότηση, όπως λέτε ο κύριο Κορνέλ. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κομισιόν χαίρεται που βλέπει το ενδιαφέρον τη Επιτροπή Μεταφορών για το θέμα αυτό. Συμφωνούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ασφάλεια στον αεροπορικό τομέα και θα συμβάλλει προφανώς σε καλύτερη προστασία των ταξιδιωτών και των Ευρωπαίων πολιτών. Η Κομισιόν θέλει να ευχαριστήσει τα μέλη της Επιτροπής σας και ιδιαίτερα στην κυρία Ντεβερά, την εισηγήτρια, γιατί οι τροπολογίες που έχουν κατατεθεί από την εισηγήτρια αλλά και από τους σκιώδεις και τα άλλα μέλη της Επιτροπής φέρνουν κάποιες αλλαγές στην, Επιτροπή, στην πρότασή μας που γενικά μπορεί να τις υποστηρίξει η Κομισιόν καθώς πηγαίνουν στην ίδια κατεύθυνση και ακολουθούν τους στόχους που έχουμε θέσει και εμείς οι ίδιοι. Τέσσερις περιπτώσεις θέλω να αναφέρω. Η Κομισιόν βλέπει πολύ θετικά τις τροπολογίες που θέλουν να ενισχύσουν τη σωστή κουλτούρα στον τομέα αυτό και την προστασία για τους επαγγελματίες του αεροπορικού κλάδου. Δεύτερον, η Κομισιόν υποστηρίζει το να έχουμε πιο αναλογικούς κανόνες σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις, <clears throat> σε ό,τι αφορά ε, τα αεροσκάφη αναψυχής και τα ελαφρά αεροσκάφη. Η Κομισιόν επίσης υποστηρίζει τις προτάσεις που έχουν σαν στόχο να ε, αντανακλάται περισσότερο ο διπλός ρόλος της ΕΑΣΑ σαν συντονιστή πρώτα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για σημαντικά θέματα ασφάλειας και δεύτερον ως αρχή πιστοποίησης ε, αντίστοιχη με αυτή των κρατών μελών στο δικό της τομέα αρμοδιότητας. Και είναι πολύ σημαντικές οι διευκρινήσεις αυτές του ρόλου της ΕΑΣΑ. Τέλος, η Κομισιόν βλέπει θετικά όλες τις συμβαστικές προτάσεις της εισηγήτριας, εκτός από την 6 για τις κατε εξουσιοδότηση πράξης και την 7 για την υποχρέωση παροχής αναφορών από την Κομισιόν. <clears throat> Πρέπει να αναφέρω κάποιες τροπολογίες που η Κομισιόν δεν μπορεί να υποστηρίξει. Πρώτα απ' όλα, η Κομισιόν δεν υποστηρίξει τις τροπολογίες 85, 88, 120, 120 142, συγγνώμη, γιατί αποδυναμώνουν την προστασία των ε, επαγγελματιών στο χώρο της αεροπορίας που δίνουν αναφορές και επομένως θα αποδυναμώσουν την σωστή κουλτούρα στον τομέα αυτό. Δεύτερον, η Κομισιόν δεν υποστηρίζει τις τοπολογίες 118 και 132 γιατί περιορίζουν την εμβέλεια των ε, συμβάντων που πρέπει να αναφέρονται. Η Κομισιόν θεωρεί ότι ο αεροπορικό κλάδο δεν θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αποκρύπτει σημαντικέ πληροφορίε από τα κράτη-μέλη και την ΕΑΣΑ. Επιπλέον η Κομισιόν δεν υποστηρίζει την τροπολογία 95 γιατί από νομική απόψη είναι αμφισβητήσιμο αν μπορεί να συμπεριληφθεί μια τέτοια διατύπωση στο άρθρο σε σχέση με το εύρο εφαρμογή, γιατί και ο βασικό κανονισμό 2.16 τη ΕΑΣΑ και αυτό ο κανονισμό έχουν διαφορετικές, διαφορετική σφαίρα εφαρμογή και επίση. Ο εφαρμοστικός κανονισμός του 216 του 2008 περιλαμβάνει την ίδια ρήτα, τις ίδιες ρήτες με την επιφύλαξη τριστελείς, όπως και εδώ. Επομένως έχουμε μια κυκλική κατά κάποιο τρόπο μορφή αναφοράς που οδηγήσει σε συγκρούσεις και νομική ανασφάλεια που θα δημιουργήσει πρόβλημα για τη σωστή εφαρμογή αυτού του νέου κανονισμού. Κατανοούμε <clears throat> το λόγο για τον οποίο κατατέθηκε αυτή η τροπολογία, αλλά θεωρούμε ότι η τροπολογία της ηγητρίας Παϊθμών 1 είναι πιο εύστοχη για να αντιμετωπίσει το θέμα αυτό της διάδρασης μεταξύ αυτού του κανονισμού αφενός και του 2.16 του 2008 με τους εφαρμοστικούς κανόνες της. Του. Τέλος η Κομισιόν θεωρεί ότι οι συμβαστικές τροπολογίες 6 και η τροπολογία 77, 87, 146, 148, 149 και 150 θα δημιουργούσαν μια διαδικασία για την εφαρμογή των κατεξουσιοδότηση πράξεων που δεν συνάδει με το άρθρο 290 των συνδικών και επίσης δεν συμφωνεί με την κοινή κατανόηση για τις κατεξουσιοδότηση εξουσίες που έχουν συμφωνήσει τα κράτη-μέλη και δεν υποστηρίζει τις τροπολογίες 96 και 156 γιατί έχουν σαν στόχο να προσθέσουν στις ε, ε, υποχρεώσει που βρίσκονται στο βασικό έγγραφο και πολλέ πρέπει να μείνουν στι και πράξη. Η Κομισιό θέλει και πάλι να ευχαριστήσει την εισηγήτρια κατά μέλη τη Επιτροπή σα για την υποστήριξη που μα έχετε δώσει, την ισχυρή υποστήριξη για τη γενική κατεύθυνση τη προτάσεώ μα και του στόχου τη Νέα αυτού κανονισμού και για το γεγονό ότι έχετε καταθέσει τροπολογίε που έχουν βελτιώσει τα μάλα αυτήν την πρόταση. Επειδή βάσει τη αυριανή ψηφοφορία νομίζω ότι μπορούν να γίνουν σημαντικέ και επιτυχής διαπραγματεύσει ώστε το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να καταλήξουν σε ένα κείμενο το οποίο θα οδηγήσει σε συγκεκριμένες ε, διατάξεις για την προστασία των πολιτών και την αναφορά αεροπορικών συμφάτων. Κύριε Ντέιβερα, θέλετε να πείτε κάτι. Oui, rapidement, euh, concernant Cassine, je, je comprends l'inquiétude qu'il Πολύ σύντομα. Ε, σε σχέση με τον κύριο Καντζέν για τις αμφιβολίες που εξέφρασε για τους μικρούς οργανισμούς, μικρές δομές και εγώ προσπάθησα να ελαφρύνω κάπως τα πράγματα και αυτό που προτείνουμε στον Συμβαστική 5 είναι ένας απλοποιημένος μηχανισμός για την ανησυχία της κυρίας Φώστερ και του κυρίου Γκράντες ε, ε, έχουμε προσεγγίσει αυτόν τον ορισμό στην 7η Συμβαστική και συνεργαστήκαμε με αστυνομική υπηρεσία και όπως είπατε κύριε Πρόεδρε και όπως είπε και η Εύα Λίχτεμπέργκερ η ε, ποινική ύλη δεν έχει ευθυγραμμιστεί δηλαδή το θέμα του δόλου ή της αμέλειας δεν είναι ομοιόμορφη. Δεν είναι ε, βέβαια εδώ καθολικός αυτός ο ορισμός, αλλά ισχύει μόνο για αυτό εδώ το κείμενο. Θέλω να σας ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω την Επιτροπή Μεταφορών και την Κομισιόν για την αλλαγή απόψεων και για τη δουλειά που κάνουμε μαζί και που μας επιτρέπει να έχουμε αυτή την έκθεση έτοιμη σήμερα. Θα ήθελα αύριο, Πρόεδρε, μετά από την ψηφοφορία να καλέσουμε τα μέλη να ψηφίσουν για μια εντολή που θα επιτρέψει την ταχύα έναρξη του τριμερού διαλόγου με στόχο να προσπαθήσουμε να έχουμε συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση στους επόμενους μήνες για να μπορέσουμε και να την υιοθετήσουμε πριν το τέλος της θητείας σας. Ευχαριστώ. Thank you very much, Mrs. Remind will be... Σας πενθυμίζω ότι ψηφίζουμε αύριο, αν θέλει ο Θεός και επίσης θα ψηφίσουμε για, με την ψηφοφορία για την εντολή διαπραγματεύσει. Ερχόμαστε τώρα στην ανάπτυξη ε, μιας υποδομής αναλλακτικών καυσίμων με τον Κάρλο Φιτάντσα ως εισηγητή. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτή η πρόταση προέρχεται από την Κομισιόν και εντάξετε στο πλαίσιο μια γενικής στρατηγική που αφορά α πούμε ε, τα ανανεώσιμε πηγέ πηγές ενέργειας. Εμείς ε, θα εξετάσουμε την οδηγία CARS 2020 και διάφορες άλλες. Η δική μου πρόταση έκθεσης ε, καταρχήν να ξεκινά από μια γενικά θετική εξέταση της θέσης που θέλησε να μας προτείνει η Κομισιόν Φυσικά προβλέπεται μια σειρά από τροπολογίες για να βελτιωθεί η πρόταση της Κομισιόν. Νομίζω πως όλοι συμμεριζόμαστε την ανάγκη και τη σημασία επένδυσης σε εναλλακτικά κάψιμα στην Ένωση για να μειώσουμε την εξάρτηση του, την εξάρτηση από το πετρέλαιο, τουλάχιστον σε οδικές μεταφορές, αλλά να μειώσουμε και την περιβαλλοντική ρήπανση και τις εκπομπές ε, ρηπογόνων αερίων. Τα πιο σημαντικά στοιχεία της έκθεσης είναι τα εξής. Ε, καταρχήν τα εθνικά ε, στρατηγικά σχέδια τα οποία μέσω εθνικών στόχων και στρατηγικών σχεδίων ανάπτυξης για την ανάπτυξη των ελεκτικών καυσίμων που προβλέπονται ως στοιχεία ε, και να τα έχουμε δηλαδή στην ημερομηνία του 2020. Δεύτερον, στρατηγική προσέγγιση που θα λαμβάνει υπόψη διάφορα είδη εναλλακτικών καυσίμων. Αρχικά το κείμενο αυτό ξεκίνησε με μια ιδιαίτερη προσοχή στην ηλεκτρισμό, ενώ στην πρόταση που προέκυψε από την Κομισιόν ε, συμπεριλήφθηκε συλλήφθηκαν εδώ όλα τα είδη εναλλακτικών καυσίμων εκτός από τα στερεά δηλαδή και προσπαθήσαμε να προβλέψουμε και το τρόπο μεταφορών που αυτή τη στιγμή για τεχνολογικούς λόγους δεν έχουν ακόμα αναπτύξει μια αξιόπιση εναλλακτική για τα ε, στερεά καύσιμα ε, όπως ας πούμε τα αεροσκάφη. Έχω ενσωματώσει εδώ και κάποιους ενδιάμεσους στόχους για να μπορούμε να παρακολουθήσουμε τα βήματα που θα κάνει κάθε χώρα τη στιγμή που θα τεθεί ενισχύ αυτή η οδηγία. Όσον αφορά τη, τα ηλεκτρικά μέσα μεταφορών υπάρχει ένας φιλόδοξος στόχος από πλευράς της Κομισιόν να προβλεφθεί δηλαδή ε, συγκεκριμένο στάνταρ για όλα τα κρατημέλη ώστε να ξεπεραστούν τα τεχνολογικά, η τεχνολογική φραγμή, δηλαδή να μπορεί να είναι εγγυημένη με τη δυνατότητα μετακίνησης ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε ένα θέμα το οποίο είναι δύσκολο να λυθεί και αφορά τον εντοπισμό ενός ενιαίου στάνταρ για τα, τις πρίζες ε, ε, σύνδεσης με το εναλλασσόμενο ηλεκτρικό ρεύμα. Και αυτό πρέπει να το δούμε και με την νομική υπηρεσία, γιατί σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες έχουμε πολύ προηγμένη ε, νομοθεσία που προβλέπει τεχνική προαπέτηση. Α, ας πούμε να υπάρχουν ρυθμιστές του ρεύματος εντός των, των εντός ε, των σταθμών ε, ε, ανεφοδιασμού. Έχουμε λοιπόν αυτή την πρόταση της Κομισιόν, αλλά προβλέπουμε εμείς και τη δυνατότητα, όταν αυτό προβλέπεται και από την νομοθεσία της κάθε χώρας, αυτές οι πρίζες δεύτερου τύπου να φέρουν διακόπτες ασφαλείας. Στα αγγλικά αυτά ονομάζονται shutter, ασφάλειες δηλαδή. Ε, εδώ δεν υπάρχει ομοφωνία ακόμα. Υπάρχει και ένα παρόμοιο θέμα που αφορά τη σύνδεση για την γρήγορη φόρτιση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων και εδώ πρέπει να βρούμε μια λύση ώστε να μπορεί να τηρείται το στάνταρ της Κομισιόν, το κόμπο 2 όπως αποκαλείται, και να συνδυάζεται με άλλες τεχνολογίες που ήδη κυκλοφορούν στην αγορά, όπως η ε, τεχνολογία σαν demo, που έχει ε, επεκταθεί αρκετά, να προβλεφθούν δηλαδή μηχανισμοί που να είναι ουδέτεροι και να μην επιβάλλουν τη χρήση της μίας ή της άλλης ε, ε, τεχνολογίας. Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα φόρτισης Wi-Fi, άνευ καλωδίων δηλαδή. Αυτή τη στιγμή αναπτύσσεται αυτή η τεχνολογία. Υπάρχει ακόμα ένα μεγάλο θέμα που αφορά το στόχος που προβλέπονται για κάθε κράτος μέλος. Εδώ υπάρχει ευρύτατη συζήτηση και στο εσωτερικό του Συμβουλίου, γιατί πολλές χώρες θεωρούν πως ε, οι στόχοι αυτοί ε, δεν ανταποκρίνονται στις εθνικές πραγματικότητες. Ε, εγώ σε σχέση με αυτό δεν έχω παρέμβει, δεν έχω αλλάξει τα νούμερα. Θεώρησα πως δεν είχαμε αρκετά τεχνικά στοιχεία στη διάθεσή μας για να μπορέσουμε να στηρίξουμε διαφορετικές ποσότητες σε σύγκριση με αυτές που υποδεικνύει η Κομισιόν και νομίζω πως κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων θα μπορέσουμε να βρούμε μια κοινή λύση. Θεωρώ ωστόσο ότι δεν θα πρέπει να κενωθεί περιεχομένου η πρόταση αυτή. Εάν προβλέπαμε ότι αυτή η στόχη, αυτό το παράρτημα θα κυρωθεί ή θα βγει από το οριστικό κείμενο ή ότι αυτή η στόχη δεν θα είναι πια δεσμευτική αλλά θα είναι ενδεικτική, στην ουσία δεν θα έχουμε λόγο να φτιάξουμε, να κάνουμε καμία εργασία. Θεωρώ λοιπόν πως είναι πιο χρήσιμο να μιλάμε για πιο συγκεκριμένες ημερομηνίε, αλλά για ομαλή προσγείωση ώστε όλες οι χώρες να μπορέσουν να πετύχουν τους προβλεπόμενους στόχους, αλλά όχι να κενώσουμε είναι οδηγία περιεχομένου. Τώρα όσον αφορά το υδρογόνο, γνωρίζουμε πως αυτό το εναλλακτικό κάψιμο δεν έχει αναπτυχθεί τόσο όσο άλλα, ακόμα και αν υπάρχουν ενδιαφέρουσες προοπτικές για βελτίωση. Εγώ έχω απλά επιβεβαιώσει τα νούμερα και τις προβλέψεις που περιλαμβάνονται στην πρόταση οδηγίας από πλευράς της Κομισιόν. Έχω ωστόσο προβλέψει να μην χρειάζεται να αναπτυχθεί το δίκτυο του υδρογόνου μόνο στα κράτη-μέλη όπου ήδη υπάρχει και όπου προβλέπεται μια προθεσμία για το 2020, αλλά θα πρέπει να γίνουν επενδύσεις και στις άλλες χώρες όπου ακόμα αυτό το κάψιμο δεν χρησιμοποιούνται τόσο προβλέποντας βέβαια μακρύτερα χρονικά περιθώρια, τα οποία έχουμε ορίσει στο 2030. Μεγάλη σημασία θέλησα να δώσω εξάλλου στο θέμα του φυσικού αερίου, τόσο συμπιδεσμένο όσο και το υγρό φυσικό αέριο. Το LNG είναι αποτελεσματική εναλλακτική όσον αφορά το κόστος και την ε, ε, οικονομία, ιδιαίτερα για τις πλωτές οδούς, ιδιαίτερα για τις μεταφορές ε, σε λάστιχο. Αντιθέτως όσον αφορά τις πλωτές οδούς και τις θαλάσσιες μεταφορές, η Κομισιόν προβλέπει σε όλα τα λιμάνια να προβλέπεται μια εγκατάσταση ανεφοδιασμού LNG. Εγώ πιστεύω πως αυτή η διάταξη είναι εξαιρετικά δεσμευτική και θα πρέπει να αφήσουμε μεγαλύτερη ελευθερία στα κρατημέλη ώστε να μπορούν να ορίσουν εντός του εθνικού τους σχεδίου ποιε λύσεις μπορούν να είναι χρήσιμες. Αν σκεφτώ α πούμε τη χώρα μου, το να προβλέψουμε στο λιμάνι τη Γένοβας και σε λίγα χιλιόμετρα στο λιμάνι τη Λασπέτσια να υπάρχουν δύο εγκαταστάσει που θα κάνουν την ίδια δουλειά, νομίζω πως είναι οικονομικά αβάσιμο, μη βιώσιμο και δεν χρειάζεται. Μεγαλύτερη ευελιξία λοιπόν σε αυτό το σημείο ζητάω και όσον αφορά το συμπιεσμένο φυσικό αέριο έχω προβλέψει να περιορίσω το minimum, την μίνιμουμ ακτίνα εγκατάστασης για το συμπιεσμένο φυσικό αέριο ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη εξάπλωση του δικτύου και υπάρχει και θέμα όσον αφορά το GPL. Γιατί η Κομισιόν προβλέπει στο κείμενό της στην εισαγωγή, στον, στον κατάλογο δηλαδή των εναλλακτικών καυσίμων, το GPL, που όμως μετά στο παράρτημα εξαφανίζεται. Δεν αναφέρονται δηλαδή πραγματικοί στόχοι. Γνωρίζουμε όμως αυτό το, το είδος του καυσίμου έχει μεγάλη διάδοση σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι της Ευρώπης. Είναι λιγότερο καθαρό από τα άλλα εναλλακτικά καύσιμα που περιλαμβάνονται στο κείμενο της οδηγίας, αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρξει μια υπόθεση ανάπτυξης και για αυτό το δίκτυο. Και κλείνω έδωσε ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα της ποιότητας των καυσίμων, πράγμα που εντάσσεται και στην εργασία που κάνουμε για άλλους κανόνες για την οδηγία για την ποιότητα των καυσίμων. Ε, επίσης δίνουμε μεγαλύτερη προσοχή στον τελικό καταναλωτή, στον πελάτη και προτείνω εναρμόνιση των χρωμάτων των αντλειών για τις διάφορες, τα διάφορα καύσιμα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει απόλυτη ομοιομορφία. Όταν αλλάζει χώρα αλλάζει και το χρώμα που... του κάθε καυσίμου στο σταθμό. Τελευταίο θέμα είναι το θέμα της χρηματοδότησης για αυτές τις επενδύσεις και αυτές τις υποδομές. Ζητήσαμε μια μελέτη και συγκεκριμένη ανάλυση από την Κομισιόν για να δούμε πώς πέρα από τις παρεμβάσεις και τις επενδύσεις από τον ιδιωτικό τομέα, είτε είναι κατασκευαστές αυτοκινήτων, είτε είναι διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, είτε άλλοι, να υπάρχει δυνατότητα να έχει κανείς πρόσβαση στα χρήματα της ε, Ευρωπαϊκής ε, Τράπεζας Επενδύσεων και άλλα ταμεία ευρωπαϊκά που να μπορούν να στηρίξουν τις προσπάθειες των κρατών μελών και των ιδιωτών για την εξάπλωση αυτών των δικτύων. Ευχαριστώ. Έχουμε 7 ομιλητές και την Κομισιόν. Παρακαλώ να είστε πολύ σύντομοι. Ήδη είναι η πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Θα έχουμε ε, συζήτηση πιο εις βάθος ε, κατά τη συζήτηση των τροπολογιών. Ο κύριος Έρτουγκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Φιντάντσα, τον εισηγητή, για την, ε, το ανοιχτό πνεύμα που έχει δείξει στη συνεργασία μεταξύ μας και για την εξισορροπημένη πρόταση ευθεσής του. Γενικά υπάρχει υποστήριξη της πρότασης της Κομισιόν και εγώ συμμεριζόμαι πάρα πολλά που, από αυτά που ανέφερε ο εισηγητής για μένα. Το πιο σημαντικό θέμα είναι πώς θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε τις εθνικές στρατηγικές. Αυτό πιστεύω ότι πρέπει να το υποστηρίξουμε αν θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να δημιουργήσει ένα ευρύ χώρο ο οποίος όμως θα έχει και την ευκαμψία να ενσωματώσει τις εθνικές ιδιαιτερότητες και να μπορέσει με λυσιτελή τρόπο να, λειτουργήσει και επίσης πιστεύω ότι ε, ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι οι ενέργειες που θα γίνουν για να υποστηρίξουμε τα διάφορα εναλλακτικά καύσιμα. Πρέπει η τεχνολογία, όπως είπε και ο εισηγητής για τα νέα αυτά καύσιμα, να αποδείξει ακόμα την αξία τους και είναι απαραίτητο να έχουμε και την έκθεση αντικτύπου της Κομισιόν που να δείξει πώς θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τα εμπόδια που υπάρχουν σε σχέση με ορισμένα ε, εναλλακτικά καύσιμα. Πιστεύω ότι τελικά θα πρέπει να υποστηρίξουμε όλο αυτό που έχουν να κάνουν με την ε, ε, επιδότηση όλων των τεχνολογιών που προωθούν το φυσικό αέριο και την ε, υδροελεκτρική ενέργεια. Σε ό,τι αφορά τώρα το υγροποιημένο φυσικό αέριο και τα βιοκαύσιμα, το, συγγνώμη, το LPG μάλλον, το φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται στα οχήματα, ξέρετε ότι αυτό είναι παραπροϊόν της παραγωγής βενζίνης και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί για την υποστήριξή του. Το απαραίτητο είναι το νομικό πλαίσιο να διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια σαφή στρατηγική και επομένως όλη αυτή η διαδικασία να ενισχυθεί και να δια... διευκολυνθεί και ενώ συγχρόνως να μπορέσουμε να αποφύγουμε λαθασμένες αντιμετωπίσεις. Πρέπει λοιπόν ένα μεγάλο μέρος αυτής της διαδικασίας να επαφείεται στα κράτη-μέλη. Τέλος, να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχουν συμβατά πρότυπα για όλες τις τεχνικές, αλλά πάντα υπάρχει η λογική των first movers, αυτοί δηλαδή οι οποίοι για πρώτη φορά ξεκινάνε σε ένα νέο τομέα, θα πρέπει <clears throat> να τους ε, ενισχύσουμε και αυτό είναι κάτι το οποίο με οδηγεί στην ανάγκη να έχουμε ένα κατάλληλο ε, πλαίσιο χρονικό για τις πρίζες, παραδείγματος χάρη, όπως ελέγχθη, για την εναρμόνισή του. Μας ενδιαφέρει επίσης να υπάρξει και φιλική προς τον καταναλωτή ετικετοποίηση για τις αντλίες ώστε να μπορεί να είναι σαφές περί τίνος πρόκειται. Και τέλος ένα ακόμα σημείο το οποίο είναι κριτικού χαρακτήρα πιστεύω είναι το θέμα της χρηματοδότησης. Ξέρουμε ότι δεν μας βγαίνουν από τα αυτιά τα χρήματα. Θα ήταν χρήσιμο εδώ τα διευρωπαϊκά δίκτυα να ενισχύσουν την ε, υποστήριξη αυτών των ε, <clears throat> εναλλακτικών καυσίμων. Αλλά αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι τα κρατημέλη έχουν επιμείνει τα χρήματα αυτά να ε, επενδυθούν περισσότερο στο σιδηρόδρομο και τις εσωτερικές υδάτινες οδούς και όχι στην οδική μεταφορά. Μάλιστα, ναι. και εγώ θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον εισηγητή. Νομίζω ότι είναι πολύ καλή αυτή η έκθεση. Αναφέρθηκε το θέμα των TNT, των διευρωπαϊκών δικτύων, όπου έχουμε λάβει υπόψη την ανάγκη να επενδύσουμε για καλύτερα διευρωπαϊκά δίκτυα για εναλλακτικές μορφές αυτοκινητοκίνησης σε ό,τι αφορά την ε, ηλεκτροκίνηση Ξέρουμε όλοι ότι πρέπει να υπάρξει μια ενιαία μορφή πρίζα στην Ευρώπη <clears throat> για τα ευρωπαϊκά ε, οχήματα. Θα ήθελα επίσης να μιλήσω και για το φυσικό αέριο. Νομίζω ότι αυτή είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να προωθήσουμε τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Αυτή τη στιγμή πάρα, πολλές, ε, πολλά βενζινάδικα λειτουργούν ε, ως υποκαταστήματα των εταιριών πετρελαίου και δεν έχουν πολύ ενδιαφέρον να προωθήσουν τα καύσιμα, τα εναλλακτικά καύσιμα. Και όπως ελέγχθη ε, από τις τροπολογίες 53 και 63 υπάρχουν και κάποιες ε, φιλόδοξες προτάσεις για να υπάρξουν και αποθηκεύσεις φυσικού αερίου, γιατί αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την πρόθεση πλοίων, το αέριο, αλλά και για τα φορτηγά. Υπάρχουν τα προβλήματα που αναφέρθηκα με το LPC, με το υγροποιημένο ε, προπάνιο. Είναι κάτι το οποίο προέρχεται ουσιαστικά από την εξόριξη πετρελαίου από την επεξεργασία καλύτερα του πετρελαίου. Αυτό δεν είναι ακριβώς μια αναλλακτική ενέργεια ή μια ανανεώσιμη <clears throat> μορφή ε, ενέργειας. Δεν είναι το ίδιο πράγμα λοιπόν με το φυσικό αέριο. Το προπάνιο, το ευρωποιημένο προπάνιο είναι λιγότερο ανανεώσιμο από το φυσικό αέριο. Δεν δίνει τις ίδιες δυνατότητες εξοικονόμησης. Και εξάλλου η υποδομή για το LPG, το υγροποιημένο προπάνιο, υπάρχει ήδη στην Ευρώπη, είναι 3.000 ε, τα βενζινάδικα που δίνουν το LPG και άλλα 3.000 για το φυσικό αέριο. Και κατανοώ αυτό που λέτε για το ότι δεν πρέπει να βρισκόνται σε μειονέκτημα τα βενζινάδικα τα οποία προσφέρουν αυτές τις νέες μορφές εναλλακτικών καυσίμων. Τέιλορ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και πάρα πολύ σύντομα γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Συμφωνώ ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση για να ε, υπάρξουν συγκεκριμένες προδιαγραφές. Αλλά ο βασικός στόχος ε, όλης αυτής της ιστορίας με τα αναλλακτικά καύσιμα είναι οι μεταφορές να ε, ε, έχουν λιγότερες εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Και αυτό το κάνουμε μεταφέροντας τις, τους επιβάτες, αν θέλετε, όχι από τα ιδιωτικά αυτοκίνητα, στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και υπάρχουν πολλές εταιρείες που ε, θα πρέπει να διαθέσουν ε, παραδείγματος χάρη ε, φυσικό αέριο στα βενζινάδικα, στους αυτοκινοδρόμους κτλ ή, ή άκουσα ότι θα υπάρξει μόνο για τις εναλλακτικές για τα μικροκαύσιμα το 1% ε, της αγοράς, άρα δεν χρειάζεται τα επομένως τα, ε, τα βεζινάδικα να, πουλάνε, να έχουν πρίζες για ηλεκτρικό ρεύμα. Τέλο πάντων, το όλο θέμα όλων των υποδομών είναι κάτι το οποίο πρέπει να ε, ρυθμίσουμε πριν ε, προχωρήσουμε περαιτέρω. Ίσως ε, τα κράτη-μέλη να βρούνε τα χρήματα μόνοι τους, αλλά εγώ πιστεύω πριν δεσμεύσουμε οποιοδήποτε δημόσιο χρήμα θα πρέπει να εξετάσουμε κατά πόσον ο στόχος, δηλαδή η μείωση εκπομπών ε, διοξιδίου του άνθρακα επιτυγχάνεται καλύτερα μέσα από αυτό τον συγκεκριμένο μηχανισμό. Θα πρέπει να επενδύσουμε ίσως περισσότερο στην έρευνα και στην ε, ανάπτυξη σαν ε, άλλη λύση εκτός από τα αναλλακτικά καύσιμα. Τέλος πάντων, ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε τη δυνατότητα να μιλήσω. Κύριε Βαντάμα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον ε, εισηγητή πιστεύω ότι ο συνάδελφός μας, κύριος Τέιλορ, ε, έθιξε την καρδιά του προβλήματος. Το στόχος μας είναι να περιορίσουμε τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο που αποτέλεσε αντικείμενο ενθουσιασμού και στο παρελθόν. Μέσα στα πλαίσια αυτού του φακέλου, του θέματος, αυτό το οποίο είναι σημαντικό είναι να τονίσουμε ε, να υπογραμμίσουμε τη σημασία αυτών των εναλλακτικών καυσίμων, όχι μόνο για τις οδικές μεταφορές ή για τις ε, και τις πλωτές μεταφορές, θα πρέπει να βελτιώσουμε, αν θέλετε, τις δυνατότητες ε, χρήσης σε όλα τα σε συνδυασμένε μεταφορές και θα πρέπει να ε, δούμε τι γίνεται και με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Προχωράνε τα πράγματα γρήγορα, υπάρχει και ιδιωτική έρευνα. Αλλά ε, είμαι, αντιμετωπίζω με κάποιο σκεπτικισμό αυτό που είπε ο εισηγητής για το υποχρεωτικό σημείο φόρτισης. Για τις πρίζες ε, ε, και για το πόσο θα γίνονται οι ενώσεις και λοιπά, αυτά, τους, οι συνδέσεις, συγγνώμη, αυτό θα πρέπει να δούμε και πώς εξελίσσεται και η αγορά. όταν μπήκαν στην αγορά όλα αυτά τα αναλλακτικά καύσιμα ε, και το ηλεκτρική ενέργεια είδαμε ότι υπήρξαν σε, σε κάποια κράτη-μέλη, εμφανίστηκαν τέτοιου είδους ε, ε, πρίζες και δυνατότητες φόρτισης. Ίσως θα πρέπει επομένω να αφήσουμε και την ιδιωτική αγορά να προχωρήσει. Το GPL είναι ένα προϊόν παράγωγο του πετρελαίου. Το έχουμε συζητήσει πολύ και εδώ δεν μπορώ να πω ότι συμφωνώ με τον εισηγητή. Η κυρία Uh, well, thank you very much, Chair, and thanks to the rapporteur. Yeah, I made a few comments on this um, initially. Ευχαριστώ. Εκτιμώ την εργασία του εισηγητή, αλλά και πάλι να μιλήσω για κάποια πράγματα. Η Κομισιόν εξέτασε τέσσερις τύπους ενέργειας και μετά θα πρέπει να δούμε στην πραγματικότητα τι είναι το καταλληλότερο για κάθε κράτος μέλος. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη, νομίζω, να αποφασίζουν τις πολιτικές τους για να μπορέσουν να επιτύχουν αυτούς τους στόχους, διότι εξαρτάται που βρίσκεται κανείς ε, γεωγραφικά. και πώς θα μπορέσεις να περιορίσεις τις εκπομπές, όπως είπε και ο κύριος, ε, ε, Τέιλορ. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Το 2020 με όλο το σεβασμό δεν νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Δεν έχει νόημα να βάζουμε τέτοιους στόχους. Είναι κάτι το αδύνατον. Τώρα, για το πώς θα πήγαινε το πράγμα, πώς ε, θα μπορούσες να κινηθείς από χώρα σε χώρα αν είχες τέτοιο αυτοκίνητο. Εσείς το αγγίξατε το θέμα εδώ, πρόκειται για μαζικές, ε, μεγάλες υποδομές που πρέπει να φτιαχτούν και η αγορά είναι αυτή που θα πρέπει να τα καθοδηγήσει όλα αυτά. Τώρα δεν ξέρω αν η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει λεφτά για να τα κάνει όλα αυτά. Εγώ είχα την εντύπωση πως αυτά τα δύο αυτοκίνητα στην πλατεία Λουξεμπούργκ είναι εκεί στην πρίζα αλλά δεν έχω δει ποτέ κανέναν να πηγαίνει να τα παίρνει, να τα οδηγεί. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Ένωση καλά να χρηματοδοτήσει ένα σωρό μπρίζες και τέτοια, αλλά η αγορά θα πρέπει να είναι κατά τη γνώμη μου αυτή που θα το κάνει, γιατί και τα κρατη δεν έχουν λεφτά. Δεν ήρθε κανένα κάτω μέλο να μα πει ε, α ξοδέψουμε μισό για να τα φτιάξουμε όλα αυτά. Ούτε έτσι λειτουργεί το πράγμα. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι πρόβλημα το να θίγουμε θέματα, ε, να δούμε πώς θα γίνουν δηλαδή, πώς θα κάνουμε αυτές τις αλλαγές που θέλουμε να κάνουμε. Το συζητάμε, ναι, αλλά ίσως θα πρέπει να δούμε και ποια είναι η πραγματικότητα και πού βρίσκονται τα κράτη-μέλη. Εγώ δεν έχω ιδέα τι κάνουν όλοι οι υπόλοιποι και τι έχουν και τι δεν έχουν. Δεν είναι αρνητική η στάση μου, απλά νομίζω πως είναι κάπως ε, υπεροπτικό ε, το να θέλουμε να δώσουμε όλες αυτές τις οδηγίες και πολύ νωρίς για να κάνουμε κάτι τέτοιο. Α, εσείς μιλήσατε, εντάξει. Ο από την... Ο κύριος Ονίδη από την ε, DG Move. Σύντομος θα είμαι. Θέλω να τονίσω την εκτίμησή μας προς τον εισηγητή και την ε, εντύπωσή μας ότι είναι υψηλής ποιότητας αυτό το σχέδιο έκθεσης. Αν μου επιτρέπετε να, κάνω, να δώσω μια απάντηση σε σχέση με τις προτάσεις του εισηγητή για να βελτιωθεί η αρχική πρόταση της Κομισιόν. Δίνουμε μεγάλη αξία στο γεγονός στο ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη έμφαση στις ε, μεταφορές με σιδηρόδρομο. Επίσης, το γεγονός ότι αναφέρθηκε και η δυνατότητα μεταφοράς ενέργειας με ασύρματα συστήματα. Επίσης, χαιρόμαστε ιδιαίτερα στην ε, έμφαση που έθεσε ο εισηγητής στα εθνικά συστήματα. Σε τελική ανάλυση, οι στόχοι που θέσαμε και το τόνισε ο εισηγητής ότι υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι. Ο εισηγητής προτείνει να αλλάξουμε κάποιους από τους στόχους που είχαμε θέσει σε επίπεδο χιλιόμετρων και απόστασης και αντίθετα να χρησιμοποιήσουμε μια μέθοδο που βασίζεται στον αριθμό των πολιτών που ζουν σε μια περιοχή. Όλες αυτές οι μέθοδοι είναι έγκυρες. Μπορούμε να δούμε λίγο πιο προσεκτικά, να δούμε στο τέλος της ημέρας τι είναι το πιο σημαντικό. Και εγώ νομίζω ότι το σημαντικό είναι να υπάρξουν τα εθνικά πλαίσια και τα εθνικά αυτά πλαίσια να έχουν τους σημαντικούς αυτούς στόχους σε σχέση με την υποδομή. <clears throat> και εδώ έρχομαι σε αυτό που είπε η κυρία Φώστερ, που έχει μεγάλο δίκιο. Δεν συζητάμε δημόσια χρηματοδότηση νέων μορφών υποδομής. Όλα θα πρέπει να γίνουν για να υπάρχει καλύτερη ευκαιρία στις δυνάμεις της αγοράς να μπορέσουν να δημιουργήσουν την υποδομή αυτή, τα σημεία ανεφοδιασμού, τα σημεία επαναφόρτισης. Αυτό όμως μας οδηγεί να προτείνουμε εθνικά πλαίσια και αυτό ήταν και κομμάτι της λογικής που περιλαμβανόταν στο σχέδιο έκθεσης του εισηγητού. Πιστεύω ότι ο εισηγητής έχει βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο αναφέρονται οι στόχοι αυτοί, ώστε να καταλήξουμε στην καλύτερη δυνατή ένδειξη προς τους επενδυτές, ώστε αυτή η υποδομή να υλοποιηθεί. Και αν χρειάζονται να υπάρχουν δημόσιες επενδύσεις, μονάχα ως συμπλήρωμα των ιδιωτικών επενδύσεων. Εν τέλει, πιστεύω ότι για τις ε, θαλάσσιες μεταφορές χρειάζεται λίγη προσοχή, λίγη επιφυλακτικότητα, αν υπάρχει ένας τομέας όπου χρειάζονται εναλλακτικές μορφές ε, κίνησης, ε, εναλλακτικά καύσιμα, είναι ο θαλάσσιος τομέας. Είπε και η κυρία ότι υπάρχουν πολλοί περιορισμοί για τον τομέα αυτό. Χρειαζόμαστε εναλλακτικά καύσιμα και αυτή τη στιγμή στον άμεσο χρονικό ορίζοντα είναι το υγροποιημένο φυσικό αέριο. Γι' αυτό η νομοθεσία θα πρέπει να ενισχυθεί σε σχέση με την ανάγκη οι κύριοι λιμένες και θα αναφερόμαστε βέβαια στους λιμένες των διευρωπαϊκών δικτύων να έχουν υποδομές οι κύριοι λιμένες αλλά εκεί που συμφωνούμε και με τον εισηγητή είναι ότι η επιλογή της τοποθεσίας <clears throat> των εγκαταστάσεων σε κάθε λιμάνι και η μορφή του σταθμού ανεφοδιασμού, επειδή έχουμε πολλές ε, δυνατότητες, είτε ε, κινητές δυνατότητες ανεφοδιασμού, είτε ε, σταθερές. Όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν επί τη βάση μιας έκθεσης αντικτύπου που πρέπει να γίνει από τις λιμενικές εθνικές αρχές. Όλα αυτά θα είναι πάρα πολύ χρήσιμα για το υγροποιημένο φυσικό αέριο. Χρειάζεται λοιπόν κάποια επιφυλακτικότητα να λάβουμε, έχουμε αναφέρει ήδη, έχουν αναφερθεί από στα τα περιβαλλοντικά προβλήματα και κατά τα άλλα δεν είναι μια πραγματικά εναλλακτική λύση και είχε τη δυνατότητα να αποδείξει την αξία του ευρωπημένο φυσικού αέριο ως εναλλακτική λύση. Στις χώρες λοιπόν όπου η πετρελαϊκές εταιρείες έχουν δώσει αυτό το καύσιμο και όταν οι καταναλωτές για το, για το προπάνιο μάλλον, το προπάνιο, τα πράγματα έχουν προχωρήσει καλά και δεν νομίζουμε ότι χρειάζεται περαιτέρω νομοθετική υποστήριξη. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Φιντάντσα, θέλετε να πείτε κάτι σύντομα, γιατί πρέπει να κάνουμε τι των συντονιστών. Eh, πάρα πολύ γρήγορα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους ε, για, την συνεισφορά τους και νομίζω ότι υπάρχει μια βάση για να έχουμε καλή συνεργασία και στο επίπεδο των τροπολογιών. Προφανώς ε, έχουμε μια κατάσταση η οποία είναι λίγο περίπλοκη και συνθετή. <coughs> θα Πρέπει να ε, καθαρίσουμε με την Κομισιό ε, τι, θα, τι γίνεται, ε, το η κότα και το αυγό. Λέμε δεν υπάρχει δίκτυο και δεν υπάρχει αγορά. Από την άλλη πλευρά λέμε δεν υπάρχει αγορά και δεν υπάρχει δίκτυο. Εδώ, με αυτή την πρόταση, κάνουμε κάτι, αποφασίσουμε κάτι σταθερό. Λέμε, ξεκινάμε την ανάπτυξη του δικτύου, έτσι ώστε να υπάρξει και μία ανάπτυξη της αγοράς. Αυτό όσον αφορά το project, το οποίο είναι το πιο σημαντικό. Απ' την άλλη πλευρά, έχουμε και την υποχρέωση να διατηρήσουμε μια κάποια ευελιξία όσον αφορά στα στρατηγικά εθνικά πλαίσια, κυρίως όσον αφορά την ναυσιπλοεία, διότι το να επενδύσουμε ε, σε αυτού του είδους ε, την τεχνολογία θα πρέπει να προβλέψουμε και ότι οι υποδομές ε, στα λιμάνια, γενικότερα ο εξοπλισμός και οι υποδομές στο, στα λιμάνια πρέπει να προσαρμόζεται με αυτού του είδους την τεχνολογία. Βέβαια θα πρέπει να γίνεται η ανάλυση αυτή σε εθνικό επίπεδο εκ των υστέρων. Εκεί θα υιοθετηθούν τα πιο αυστηρά μέτρα. Από την άλλη πλευρά πρέπει να παρακολουθούμε την πρόταση αυτή όσον αφορά τις τεχνολογικές εξελίξεις, διότι θα πρέπει να δούμε πώς θα βελτιωθούν τα επόμενα χρόνια οι εναλλακτικές, ε, τα εναλλακτικά καύσιμα, οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας κτλ. Ε, παραδείγματος χάρη, με βάση τις ε, εμπειρίες που έχουμε στην αυσιπλοεία στη Βαλτική που χρησιμοποιούν τώρα θάνιο για τις σαν καύσιμο για τις μεταφορές. Αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται τώρα στην πρόταση της Κομισιό, αλλά χρησιμοποιείται. Άρα για αυτό το λόγο θα πρέπει να έχουμε ανοιχτά, το, ανοιχτά τα μάτια μας για να ε, παρακολουθούμε και τις ε, εξελίξεις. Τώρα, όσον αφορά τους πόρους, και τελειώνω εδώ, δεν θα πρέπει να μιλάμε απλώς και μόνο για ε, άμεση χρηματοδότηση, δημόσια χρηματοδότηση, έτσι όπως αναφέρθηκε η Κομισιό, αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε ότι και σε τοπικό επίπεδο υπάρχουν διάφορα εργαλεία που θα μπορούσαν να ευνοήσουν την δημιουργία δικτύων ηλεκτρικού παραδείγματο χάρη. Αναφέρομαι στα, στις οικοδομές ή σε κάποια άλλα κίνητρα τα οποία μπορούν να επιτυχθούν σε τοπικό επίπεδο έτσι ώστε να υπάρξει μια φοροαπαλλαγή για τις ιδιωτικές επενδύσεις. ευχαριστώ. Λοιπόν, 1η Οκτωβρίου η προθεσμία για την υποβολή των τροπολογιών και ίσως ε, τα μέλη θα θέλανε να ε, δούνε ε, να διαβάσουν αυτό το φυλάδιο εδώ εάν το απαιτείτε, αν το χρειάζεστε τέλος πάντων, να έχετε όλα τα στοιχεία στο φυλάδιο εδώ, έχετε την έκθεση του κύριου Φιντάντσα, η οποία θα καλυφθεί από αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εδώ τελειώνει η συνεδρίασή μας. Ε, αύριο να σας υπενθυμίσω ότι πρέπει να φέρετε τις κάρτες σας για να ψηφίσουμε και τώρα συνεχίζουν οι συντονιστές. Καλό σας βράδυ.